Άρχεται η συνεδρίαση. Signori ε, Χτες ε, το Βρετανικό Κοινοβούλιο εξεφράστη με πολύ μεγάλη πλειοψηφία εναντίον της συμφωνίας η οποία ήταν το αντικείμενο διαπραγμάτευσης τα τελευταία δύο χρόνια με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς θα λάβουμε υπόψη μας το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αυτής με μια κάποια πικρία, αλλά φυσικά θα το σεβαστούμε, διότι είναι η έκφραση της πλειοψηφίας των πολιτικών δυνάμεων που ήσαν παρούσες στην Κάτω Βουλή. Δεν ε, διαφεύγει ότι υπάρχουν πολλές πολιτικές ε, δυνάμεις που καταψήφισαν την συμφωνία, αλλά για διαφορετικούς λόγους άλλοι ανήσυχοι για το backstop, άλλοι ευχόμενοι στενότερη σχέση με την Ένωση στο μέλλον, την διατήρηση της Τελωνιακής Ένωσης. Είναι σαφές ότι είναι νωρίς για να αξιολογήσουμε τις συνέπειες αυτής της ψηφοφορίας. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε όμως τις εξελίξεις και στο Westminster δεν υπάρχουν πλειοψηφίες υπέρ της μίας ή της άλλης υπόθεσης. διαμορφώνονται ουσιαστικά δύο αρνητικές πλειοψηφίες, μία εναντίον της συμφωνίας και η άλλη εναντίον της εξόδου χωρίς συμφωνία, αλλά δεν υπάρχει κάποια θετική πλειοψηφία. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα γίνουν προσπάθειες έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια πλειοψηφία υπέρ μιας κοινή λύσης και θα αναμένουμε για να δούμε πώς η Βρετανική κυβέρνηση θα συνεχίσει από εδώ και πέρα. Εμείς από πλευράς μας θέλουμε να επιμείνουμε στις στενές σχέσεις μας με το Ηνωμένο Βασίλειο, εφόσον το επιθυμεί και το ίδιο, και εφόσον αποφασίσει να τροποποιήσει τις κόκκινες γραμμές τις οποίες μας είχε επιβάλει. Εμείς έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στο διαπραγματευτή μας, τον κύριο Μισελ Μπαρνιέ, ο οποίος με ευφυΐα, ικανότητα και σοφία διεύθυνε και κατήφθηνε τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι τώρα αν δεν είναι δυνατόν να είμαστε όσο φιλόδεξοι επιθυμούμε, θα οδεύσουμε σε μία έξοδο χωρίς πρώτερη συμφωνία, κάτι το οποίο θα είναι αρνητικό για όλους και το παραδέχονται αυτό όλοι. Παρ' όλα αυτά θα επιταχύνουμε τις προετοιμασίες έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για μία έξοδο άνευ συμφωνίας. και αυτή είναι και η γραμμή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να μην αδικήσουμε τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο και τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει να υποφέρουν και δεν θα πρέπει να είναι τα πρώτα θύματα μιας άνευ πρώτερης συμφωνίας εξόδου. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη προσοχή το Ιρλανδικό πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουμε την Ιρλανδία. Θα πρέπει τα σύνορα ανάμεσα στη Βόρεια Ιρλανδία και την Δημοκρατία της Ιρλανδίας να είναι ένα ευέλικτο σύνολο σύνορων και να καλύπτει τα συμφέροντα της υγείας, της γεωργίας και της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Θα πρέπει να συνεχίσουμε στα πλαίσια αυτού του καθεστώτος την ενότητα των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που ε, διαμορφώσαμε κατά τη διάρκεια αυτών των μακρόχρονων και δύσκολων διαπραγματεύσεων. Μια ενότητα η οποία δείχνει ότι μπροστά στις δύσκολες καταστάσεις υπάρχει και είμαστε ικανοί να έχουμε μια συνεκτική πολιτική γραμμή. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα πλέον την συζήτηση με τις δηλώσεις της, ε, του Συμβουλίου και της Επιτροπής εξ του Συμβουλίου. Τον λόγο έχει η Υπουργός κυρία Μελάνια Τσότ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, τον Νοέμβριο πέρσι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την Συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρατόμ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την πολιτική δήλωση η οποία έθετε το πλαίσιο για τις μελλοντικές σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ηνωμένο Βασίλειο και επανέλαβε την αποφασιστικότητα της Ένωσης να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο στο μέλλον. Αυτό το αποτέλεσμα δεν θα ήταν δυνατόν χωρίς ε, την ενότητα και την υπευθυνότητα μεταξύ των 27 κρατών μελών, όπως και μεταξύ των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα, αφού μάθαμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, δεν μπορούμε παρά να λυπηθούμε για ε, το, αυτό το αποτέλεσμα και θα έχουμε μια άτακτη έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου. Μάλλον ένα τέτοιο σενάριο θα έχει σοβαρές επιπτώσεις για όλους μας, αλλά κυρίως για το Ηνωμένο Βασίλειο. Με τις τα αποτελέσματα θα πρέπει ε, να κάνουμε έκκληση για μεγαλύτερη ενότητα και υπευθυνότητα μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λόγω των πολλών ε, δισταμένων ε, σημάτων που είχαμε πριν από την συζήτηση που οδήγησε στην ψηφοφορία σε όλο το φάσμα το πολιτικό του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε μια εξήγηση γι' αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό το αποτέλεσμα βεβαίως δεν είναι το τέλος του παιχνιδιού, ενώ έχουμε ε, τα ορισμένα μέτρα. Δεν έχουμε θέμα επαναδιαπραγμάτευσης. Θα πρέπει να δράσουμε όταν το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει διευκρινίσει τι σημαίνει το αποτέλεσμα αυτό για τη διαδικασία κύρωσης και ποιες θα είναι τα επόμενα μέτρα. Εν τω μεταξύ, όπως έκανα έκκληση και έκανε έκκληση το Συμβούλιο στην πρόσκληση στην Κομισιό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα. Εξακολουθούμε την διαδικασία κύρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άποψη αυτή χαίρομαι που μπορώ να αναφέρω ότι την περασμένη εβδομάδα ήδη το Συμβούλιο υιοθέτησε την απόφαση για την υπογραφή της συμφωνίας και ενέκρινε την πρόταση αυτή όπως και ε, το αίτημα για την συγκατάθεση του Κοινοβουλίου. Η υπευθυνότητα για να εξασφαλίσουμε την κύρωση παραμένει ε, στα χέρια της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Η αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε θα έπρεπε να στηρίξει το, την κυβέρνηση για να εκπληρώσει το τελικό αποτέλεσμα ως προς το χρόνο και το περιεχόμενο Παρόλα αυτά δεν είναι βέβαιο το αποτέλεσμα. Εμείς συνεπώς πρέπει να συνεχίσουμε την προετοιμασία μας για όλες τα ενδεχόμενα ακόμα ε, και για μη συμφωνία. Δεν θέλουμε μια τέτοια κατάσταση, αλλά θα πρέπει να προετοιμαστούμε δεόντως αν υπάρξει μια τέτοια λύση. Η ετοιμότητα και ε, το έκτακτο σχέδιο ανάγκης ε, θα πρέπει να κατέχουν μεγαλύτερη σημασία εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να προετοιμαστούμε. Αυτό σημαίνει πρόσθετη νομοθετική εργασία σε αυτήν ε, την, την τελευταία φάση, αλλά έχουμε εμπιστοσύνη ότι το Ευρωπαϊκό ε, κοινοβούλιο θα ανταποκριθεί στην ε, πρόκληση όλων των ενδιαφερομένων. Το Προεδρείο με τη δική σας συνεργασία πάντως είναι αποφασισμένο να διευκολύνει την έγκριση των μέτρων εκτακτής ανάγκης εν ευθέτω χρόνο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Το λόγο έχει ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φραντς Τίμερμανς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ψηφοφορία στο βράδυ στη Βουλή των Κοινοτήτων ήταν σαφής, απορρίφθηκε η συμφωνία. η Επιτροπή λυπάται ιδιαίτερα για αυτό το αποτέλεσμα, γιατί θεωρούμε ότι ήταν ε, η καλύτερη δυνατή κατάληξη. Είχαμε δύο πλευρές που διαπραγματεύονταν, ο καθένας προσπαθούσε να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά του. Ο Μισελ Μπαρνιέ από πλευρά τη Επιτροπή έκανε μια καταπληκτική δουλειά για να διαπραγματευτεί από πλευρά των 27. Η Βρετανική κυβέρνηση βεβαίω διαπραγματεύτηκε από πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου. Και θεωρούμε ότι το αποτέλεσμα αυτή τη διαπραγμάτευση οδήγησε σε μια συμφωνία αποχώρηση που έκανε τη μικρότερη δυνατή ζημιά. Και να μην έχουμε καμία αυταπάτη το Brexit θα θίξει το Ηνωμένο Βασίλειο, θα θίξει και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ως πολιτική πρέπει να περιορίσουμε την ζημία αυτή στο μέγιστο. Και θεωρούμε ότι η συμφωνία αποχώρησης μας βοήθησε. Θα βοηθούσε προς αυτήν την κατεύθυνση. Βέβαια τώρα εμείς δεν ξέρουμε τι είδου Brexit θα έχουμε. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στην Βουλή των Κοινοτήτων, να δούμε ποια θα είναι η θέση της Βρετανικής κυβέρνησης του Βρετανικού Κοινοβουλίου και θα δούμε μετά τι θα κάνουμε. Αλλά έχουμε υποχρέωση να είμαστε προετοιμασμένοι για οποιαδήποτε δυνατή κατάληξη. Ακόμη και μία άτακτη έξοδο σε περίπτωση έλλειψη συμφωνία που θα έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις και για τον Ομένο Βασίλειο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι προετοιμασμένη για να αντιδράσουμε όσο καλύτερα γίνεται σε οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Όπως είπε και εκπρόσωπος του Συμβουλίου, θα συνεχίσουμε τη διαδικασία επικύρωσης της συμφωνίας αποχώρησης εφόσον συμφωνήθηκε. Είναι κατά τη γνώμη μας η καλύτερη κατάληξη για να υπάρξει συντεταγμένη αποχώρηση. Και να αναφέρω κάτι, μια παράθεση από το C.S. Lewis. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε και να αλλάξουμε την αρχή, αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε από εδώ που ε, είμαστε και να αλλάξουμε την κατάληξη. Ευχαριστώ πολύ. Τον λόγο έχει τώρα ο υπεύθυνο διαπραγματευτή από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, του συνόλου τη Ένωση, ο κ. Μισελ Μπαρνιέ. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, μέλη του Κοινοβουλίου, κύριε Αντιπρόεδρε, κυρία Υπουργέ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της την ψηφοφορία στην Κάτω Βουλή που έγινε χθε το απόγευμα και όπως είπε ο πρώτος αντιπρόεδρος ο κύριος Τίμερμανς η Κάτω Βουλή ψήφισε χθε με μια ξεκάθαρη πλειοψηφία, ισχυρή πλειοψηφία εναντίον της συμφωνίας την οποία είχαμε συμφωνήσει Συμβούλιο με την Βρετανική Κυβέρνηση ήδη από τον μήνα Νοέμβριο και την οποία σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχατε δεχθεί ευνοϊκά. Βέβαια τη στιγμή αυτή είναι πρόωρο να αξιολογήσουμε τις συνέπειες της ψήφου αυτής. Εμείς σεβόμεθα την ψήφο αυτή και θα συνεχίσουμε να σεβόμεθα την δημοκρατική συζήτηση στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν θα ήθελα τώρα να κάνω προφητείες για τα διάφορα σενάρια. Αυτό το οποίο έδειξε η χθεσινή ψηφοφορία είναι ότι οι πολιτικές συνθήκες και προϋποθέσεις για την επικύρωση της συμφωνίας δεν υπάρχουν στο Λονδίνο. Ε, εκφράζουμε τη λύπη μας για την ψηφοφορία αυτή, για το αποτέλεσμα αυτό, όπως το είπε και ο πρόεδρος Γιούνκερ. Αυτό είναι κάτι το οποίο συνδέεται και με την τεράστια προσπάθεια την οποία έχουμε κάνει μαζί σας και με την υπεύθυνη ομάδα ε, για το Brexit εδώ και δύο χρόνια και τη συζήτηση με, το Βρετανικό, με τη Βρετανική πλευρά, τη Βρετανική κυβέρνηση, η οποία βασίστηκε στις κόκκινες γραμμές της ίδιας της κυβέρνησης αυτής. Λυπούμεθα λοιπόν για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αυτής. Θυμίζω ότι εμείς δημιουργήσαμε από κοινού με τους Βρετανούς, με τη Βρετανική κυβέρνηση, την Συμφωνία Αποχώρησης επί μιας αντικειμενικής βάσεως λαμβάνοντας υπόψη ε, την κατανομή των συμφερόντων για να μην υπάρχουν σύνορα στην Ιρλανδία, σεβόμεθη φυσικά την επιθυμία των Βρετανών να διατηρήσουν την εθνική τους κυριαρχία στο σύνολο του εδάφους τους και συνεργαζόμενοι ε, με την, Ευρωπαϊκή, με την Βρετανική κυβέρνηση έτσι ώστε να διαμορφώσουμε το πλαίσιο μιας μελλοντική λύσεως η οποία να μην είναι μακρινή στο μέλλον και ταυτόχρονα όμως να είναι και αρκετά φιλόδοξοι όσο θα το επιτρέψουν τουλάχιστον οι βρετανικέ κόκκινες γραμμές. Διαπιστώνουμε κυρίες και κύριοι ακούγοντα τις δημόσιες δηλώσεις ότι οι βουλευτές της Κάτω Βουλής οι οποίοι καταψήφισαν την συμφωνία που έγινε αντικείμενο διαπραγμάτευσης όπως το θύμισε και ο πρόεδρός σας το έκαναν για εντελώς διαφορετικούς λόγους. Πολλές φορές πλήρως αντιτιθέμενους και αντιφατικούς ψηφοφορία αυτή, αντικειμενικά λοιπόν, δεν είναι η έκφραση μιας λεγόμενης θετικής πλειοψηφίας, η οποία θα έθετε μια εναλλακτική πρόταση στη συμφωνία που έχουμε ήδη καταθέσει. Και στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε και πολύ σωστά ο κύριος Τίμερμανς, ανήκει στις Βρετανικές αρχές να αξιολογήσουν την ψηφοφορία αυτή και η Βετανική κυβέρνηση θα πρέπει να μας πει το πώς θέλει να συνεχίσει από εδώ και πέρα προς μια διατεταγμένη αποχώρηση στις 29 Μαρτίου όπως το υπενθύμησε και ο Ντόναλτ Τάσκ χτες το βράδυ, ο πρόεδρος του Συμβουλίου. Κυρίες και κύριοι, αντίθετα από αυτά τα οποία ακούστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες και τις τελευταίες ημέρες, η συμφωνία στην οποία έχουμε καταλήξει με τη Βρετανική κυβέρνηση, μια συμφωνία 600 σελίδων, είναι μια καλή συμφωνία είναι φυσικά αποτέλεσμα ενός συμβιβασμού, αλλά είναι ο καλύτερος δυνατός συμβιβασμός. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να εργαζόμαστε με αντικειμενικότητα. Η συμφωνία αυτή παρέχει νομική ασφάλεια, ασφάλεια δικαίου, εκεί όπου το Brexit δημιουργεί ανασφάλεια όπως και κάθε διαζύγιο. Ασφάλεια για τους πολίτες και τους Βρετανούς πολίτες ε, και τους πολίτες των υπόλοιπων 27 χωρών, των οποίων τα δικαιώματα γίνονται αντικείμενο εγγύησης διαρκούς. Αυτή ήταν η βασική μας προτεραιότητα, αυτή ήταν η δική σας προτεραιότητα στο Κοινοβούλιο και η προστασία των δικαιωμάτων αυτών θα παραμείνει η προτεραιότητά μας ανεξαρτήτως των εξελίξεων ασφάλεια επίσης και για τους επιχειρηματίες και σε επίπεδο ιδιωτικό και σε επίπεδο δημόσιο όσοι χρησιμοποιούν τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και τροφοδοτούνται από αυτόν είτε είναι Βρετανοί είτε από τις υπόλοιπες 27 χώρες όλα αυτά τα προγράμματα γίνονται σεβαστά με βάση αυτή τη συμφωνία. Ασφάλεια και σταθερότητα για τη δημοκρατία της Ιρλανδίας και τη Βόρεια Ιρλανδία όπου η επιστροφή των σκληρών συνόρων μπορούμε να την αποτρέψουμε με μια ευέλικτη λύση που θα επιτρέψει και θα σέβεται το σεβασμό της κυριαρχίας του Ηνωμένου Βασιλείου και τις ελευθερίες της ενίας αγοράς στα πλαίσια της συμφωνίας του Μπέλφαστ, της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής. Και γι' αυτό ακριβώς εμείς το backstop το οποίο συμφωνήσαμε με το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να παραμείνει ένα αξιόπιστο backstop Πρέπει ένα πραγματικά αξιόπιο backstop, επαναλαμβάνει στην Αγγλική ο κύριος Μπαρνιέ. Δημιουργεί ασφάλεια για τις επιχειρήσεις και για τις δημόσιες διοικήσεις που θα έχουν στη διάθεσή τους ε, μια μεταβατική περίοδο ε, τον οποίο η μοναδική βάση βέβαια λειτουργίας θα είναι η ενδιάμεση συμφωνία η οποία θα τους δώσει χρόνο για να προετοιμαστούν και να προσαρμοστούν. Η συμβιβαστική αυτή πρόταση μας δίνει επίσης μέσω αυτής της μεταβατικής περίοδου τον χρόνο ο οποίος απαιτείται για να διαπραγματευτούμε τις μελλοντικέ μας σχέσεις επί τη βάση των πολιτικών συμφωνιών στις οποίες καταλήξαμε Ένωση και Βρετανική κυβέρνηση και κάποιες αξιολογήσεις κοινέ πολιτικές οι οποίες αφήνουν ανοιχτές τις επιλογές σεβόμενοι όμως τις βασικές αρχές των ΜΕΝ και των ΔΕΚ. Όπως και να έχουν τα πράγματα, η επικύρωση συγγνώμη, αυτής της συμφωνίας είναι απαραίτητη, είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ μας στα πλαίσια της προοπτικής της δεύτερης διαπραγμάτευσης η οποία θα πρέπει να ξεκινήσει το ταχύτερο δυνατόν σχετικά με τις μελλοντικές μας σχέσεις. Για αυτές τις σχέσεις, τις μελλοντικέ σχέσεις, αυτό που είναι το πιο σημαντικό για το μέλλον και του Ηνωμένου Βασιλείου και της Υπήρου μας, να θυμίσω ότι το κοινοβούλιο σας, το Συμβούλιο ομόφωνα, πάντα έλεγαν και λέγουν ότι εάν το Ηνωμένο Βασίλειο αποφασίσει να αλλάξει τις κόκκινες γραμμές του στο μέλλον και αν το Ηνωμένο Βασίλειο κάνει την επιλογή να σταθεί πιο φιλόδοξα και να ξεπεράσει μια απλή συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών που και αυτή είναι βέβαια σημαντική τότε σε αυτή την περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πάντα δεκτική έτσι ώστε να συνοδεύσει τις εξελίξεις αυτές και να ανταποκριθεί σε αυτές τις εξελίξεις θετικά. Αναφερόμενο στις μελλοντικέ σχέσεις, δεν αναφέρομαι στις οικονομικές εμπορικές σχέσεις, στις συναλλαγές που είναι φυσικά τόσο σημαντικές για την ανάπτυξη και τη θέση απασχόλησης σε μας. Αναφέρομαι και σε τομιακές συνεργασίες, στις οποίες εμένουν πολλές κοινοβουλευτικές ε, επιτροπές σας, πανεπιστήμια, έρευνα, αλληλεία, αερομεταφορές, μεταφορές γενικότερα, συνεργασία σε επίπεδο αστυνομικής, ε, αστυνομικού επίπεδου, δικαστικού επίπεδου, πολύ σημαντικό μετά τον Brexit, η σταθερότητα της Υπήρου μας, η ασφάλεια της Υπήρου μας, η ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου, μεγάλης χώρας, μέλους του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών, χώρα φίλη, χώρα σύμμαχος, χώρα που θα παραμείνει σημαντικό εταίρο σε ό,τι έχει σχέση με την εξωτερική πολιτική, με την ανάπτυξη της συνεργασίας στον τομέα της άμυνας. Κυρίε και κύριοι, έχουμε διεξάγει τους τελευταίους 18 μήνες μια συλλογική προσπάθεια. Η συλλογική προσπάθεια αυτή έχει επικυρωθεί σε κάθε κομβική στιγμή από την Βρετανική κυβέρνηση, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και από εσάς τους ιδίους. Νομίζω ότι θα υπάρξει λύση σε αυτό το αδιέξοδο, αλλά δεν θα υπάρξει λύση αυτή όσο δεν διευκρονιστούν οι όροι της εξόδου και δεν κατοχυρωθούν από μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία στο Ηνωμένο Βασίλειο. και γι' αυτό τα επόμενα στάδια θα πρέπει πλέον να καθοριστούν πλήρως από πλευρά της Βρετανικής κυβέρνησης. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ένα διατεταγμένο Brexit παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά μας για τις επόμενες εβδομάδες. Όμω, τη στιγμή που σας ομιλώ, κανένα σενάριο δεν μπορεί να αποκλειστεί. Και αυτό ισχύει επίσης και για το σενάριο το οποίο πάντα θελήσαμε να αποτρέψουμε. Το λεγόμενο no deal, μη συμφωνία. Είμαστε στις 16 Ιανουαρίου 10 εβδομάδε μόνο πριν το τέλο του Μαρτίου, δηλαδή τη στιγμή που επέλεξε η ίδια η Βρετανική κυβέρνηση, επέλεξε η ίδια Βρετανική κυβέρνηση έτσι ώστε να καταστεί τρίτη χώρα. 10 εβδομάδε πριν λοιπόν ποτέ ο κίνδυνο ενό no deal δεν ήταν τόσο υψηλό. Εμείς σαν βασικό στόχο έχουμε να αποφύγουμε ένα τέτοιο σενάριο. Έχουμε όμως την ευθύνη να βλέπουμε τα πράγματα ξεκάθαρα και γι' αυτό από δική μας πλευράς θα εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειες για να είμαστε προετοιμασμένοι και για αυτό το σενάριο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, εδώ και πολλούς μήνες συνεργαζόμενοι με τα κράτη-μέλη και μαζί σας, ε, πρέπει να επιταχύνουμε τις προσπάθειες αυτές, συνεργασία με όλους τους εμπλεκομένους, μέσα σε σύντομες χρονικές προθεσμίες μπορεί να κληθείτε να πάρετε μέτρα κατεπήγοντα έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες αυτού του σενάριου του απευκταίου. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας. Η πεποίθησή μας, όπως το υπενθύμησε ο Αντιπρόεδρος Τίμερμαν, είναι ότι η συμβιβαστική λύση την οποία προτείναμε μετά από 18 μήνες διαπραγματεύσεων με τη Βρετανική κυβέρνηση είναι η καλύτερη δυνατή συμβιβαστική λύση. Είναι καρπός επικοδομητικών προσπαθειών από πλευράς των δύο, των δύο μερών καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Είναι επίσης αποτέλεσμα μιας επικοδομητικής στάσης δική μα δικής μου, στα πλαίσια ηρεμίας, γαλήνης, διαλόγου και διαφάνεια. Τώρα η Βρετανική πλευρά θα πρέπει να διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίο θέλει να προχωρήσει από εδώ και πέρα για να περάσουμε στην απόσυρση τη διατεταγμένη την οποία έχει επιθυμήσει και πως πέραν αυτής της αποχωρήσεως θα οικοδομήσει μαζί μας μια εταιρική σχέση διαρκή και αποτελεσματική. Κύριε Μπαρνιέ, εγώ μπορώ ήδη να προβλέψω ότι θα έχετε την εμπιστοσύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά ήταν σαφή και μέσω του χειροκροτήματο. Σα ευχαριστώ πολύ. Και θέλω να ευχαριστήσω και την ομάδα εργασία μα που συνεργάστηκε πολύ στενά με τον κύριο Μπαρνιέ για να έχουμε την ε, βέλτιστη λύση. Και ιδιαίτερα τον επικεφαλή τη ε, ομάδα του Κοινοβουλίου, τον κύριο Φερχόφστατ, αλλά και τα άλλα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εργάστηκαν τόσο σκληρά για το θέμα αυτό. Και τώρα έχουμε τις ομιλίες. Πρώτα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Μισελ, κύριε Αντιπρόεδρε, Προεδρία του Συμβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι. Τέσσερι σύντομε παρατηρήσει. Πρώτα απ' όλα είμαι περήφανο ω Ευρωπαίο. Θυμάμαι αυτά που είχαν υποθεί πριν από δυόμιση χρόνια. Πολλοί έλεγαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ε, αντιμετωπίσει ένα φαινόμενο ντόμινο και άλλοι θα σηκωθούν να φύγουν. Θυμηθείτε όμω τώρα τι έγινε. τα 27 κράτη-μέλη είναι ενωμένα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει τι θέσει μα, Όλοι ξέρουμε τι θέλουμε. Νομίζω ότι ε, όλοι στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται την ισχύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδιαίτερα οι Ιρλανδοί φίλοι μα. Μπορούμε να είμαστε περήφανοι για αυτό που επιτύχαμε του τελευταίου μήνε, χάρη στο Μισελ, χάρη στην εργασία του και στην δέσμευση του Ζαν Κλοντ Όλα αυτά είναι πολύ καλά. Δεύτερον, 28 κυβερνήσει επιβεβαίωσαν σε τη συνθήκη και τα τρία θεσμικά όργανα είπαν αυτή είναι μια καλή συμφωνία. Και υπάρχει όμως τώρα το όχι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με σαφή πλειοψηφία Άρα οι Βρετανοί φίλοι μας θα πρέπει να κάνουν τα περαιτέρω βήματα. Υπάρχουν αυτοί που θέλουν να αποχωρήσουν ε, χωρίς συμφωνία, υπάρχουν αυτοί που θέλουν σε τα συν, αυτοί που θέλουν να παραμείνουν. Πείτε μας παρακαλώ, τι θέλετε να επιτύχετε. Δώστε μας μια σαφή κατεύθυνση. Και η Ευρώπη είναι διατεθειμένη να ολοκληρώσει τις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τρίτον, ξανασκεφτείτε τους στόχους μας. Ε, θα είναι δύσκολη η πολιτική κατάσταση στο μέλλον. Είχαμε σαφείς αρχέ, όταν ξεκινήσαμε τη συζήτηση. Για μένα, για παράδειγμα, η ιδέα τη ενιαία αγορά και τη ελεύθερη κυκλοφορία των Ευρωπαίων στην Ήπειρο, ότι μπορούν να αποφασίσουν πού θέλουν να διαμένουν. Αυτό είναι ένα τεράστιο επίτευγμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και, όπω και στο παρελθόν, θα υπερασπιστώ αυτή την αρχή. Οποιοδήποτε το αποτέλεσμα τη διαδικασία εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου. Και υπάρχουν και άλλα θέματα δεν θέλουμε να υπάρχουν έλεγχοι στην, στα σύνορα της Ιρλανδίας ή να διατηρηθούν τα δικαιώματα των ε, πολιτών. Δεν βλέπω να υπάρχει καμία δυνατότητα ελιγμών για αναδιαπραγμάτευση. Αν έχουν ε, περαιτέρω αιτήματα, τότε έχουμε και εμείς ε, το δικαίωμα να προβάλλουμε περαιτέρω αιτήματα και όλα θα ξαναρχίσουν. Θα ξανανοίξει η συζήτηση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν υπάρχει καμία δυνατότητα αναδιαπραγμάτευσης. Και τέλος, ταξιδεύω παντού στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή ως υποψήφιος, όπως ε, και πολλοί από εσά. Και δεν βλέπω κανένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θεωρεί ότι η Βρετανική προσέγγιση είναι ευφύη. Κανείς δεν μου λέει κάτι τέτοιο. Οι πολίτες της Ένωσης μου λένε ότι βλέπουν ε, πολιτικό χάο, βλέπουν οικονομική αβεβαιότητα. Γι' αυτό το κύριο μήνυμά μα στην προεκλογική εκστρατεία είναι μην ακούτε τους εθνικιστές, τους εγωιστές, είναι ψεύτες. Πολύ καλύτερα να μεταρρυθμίσουμε την Ένωση παρά να φεύγει κανείς για να επιχειρεί να καταστρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη, εξ ονόματος της Προεδρευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μετά από δύο μήνες αναβολών γνωρίζουμε τη θέση πλέον της, της Βρετανικής Βουλής. Μια τεράστια πλειοψηφία καταψήφισε την Συμφωνία Απόσυρσης και την πολιτική δήλωση που τη συνοδεύει. Είναι μια ιστορική ήττα για τη Βρετανική κυβέρνηση και την Πρωθυπουργό Μέη. Γνωρίζουμε τώρα αυτό που δεν θέλει το Βρετανικό Κοινοβούλιο αλλά 70 μέρες πριν από την τελική ημερομηνία δεν ξέρουμε το τι θέλει το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο ξεκαθάρισε την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα αρνηθεί ένα σενάριο μη συμφωνία, ένα no deal, γιατί αυτό είναι το χειρότερο σενάριο για όλους και για το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο κυρίω. Εμείς επαναλαμβάνουμε λοιπόν την δήλωσή μας αυτή, δεν αποσύρουμε, δεν ε, δεν θέλουμε να καταστήσουμε πιο χαλαρή τη συμφωνία αυτή, θέλουμε να προστατεύσουμε την κατάσταση στην Ιρλανδία και στη Βόρεια Ιρλανδία, θέλουμε να αποφύγουμε τα σκληρά σύνορα, θέλουμε να διατηρήσουμε την ενιαία αγορά, όλα αυτά δεν τα διαπραγματευόμεθα. Το να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η βασική μας προτεραιότητα και η αδίποτε λύση που απειλεί τα δικαιώματα αυτά δεν θα γίνει δεκτή. Η ασφάλεια των συνόρων είναι εξίσου σημαντική με τα επίπεδα τα κοινωνικά, τα οικονομικά, τα φορολογικά, την ισορροπία δικαιωμάτων και καθηκόντων, όλα αυτά σε καμία περίπτωση δεν θα αμφισβητηθούν. Και δεν θα υποκύψουμε επίσης σε οποιαδήποτε πρόκληση για διμερείς λύσεις, η οποία δεν θα είναι ωφέλιμη για τις δύο πλευρές η ενότητα ανάμεσα στα όργανα, η ενότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα πλαίσια της στήριξης του κύριου διαπραγματευτή μας, ήταν και θα παραμείνει η βασική μας ισχύς. Ε, είμαστε ενωμένοι και θα συνεχίσουμε να σε υποστηρίζουμε, Μισελ. Πού θα πάμε από εδώ και πέρα. Απαιτείται μια θετική πλειοψηφία από πλευρά Βρετανών. Απαιτείται ένας ξεκάθαρος ορίζοντας και μια ικανότητα να καταλήξουμε σε λύσεις. Η ψηφοφορία χθε απέδειξε ότι κάτι τέτοιο δεν υπάρχει σήμερα. Η υποστήριξη ε, από την πλειοψηφία λοιπόν της κυβέρνησης αυτής μπορεί σήμερα να την διατηρήσει στην εξουσία στην απογευματινή ψηφοφορία. Αλλά δεν δίνει την απάντηση στο σημαντικό ερώτημα ε, ή θα υπάρξει μια θετική πλειοψηφία υπέρ του Brexit και θα διαμορφωθεί στην Βρετανική Βουλή ή θα πρέπει να ξαναυπάρξει ένα δημοψήφισμα. Αν το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να αλλάξει τις ε, ερυθρές γραμμές της, ε, τότε εμείς θα παραμείνουμε ε, σε στενή σχέση μαζί του. Εμείς βέβαια τις γραμμές αυτές προσπαθήσαμε να τις συζητήσουμε, αλλά δεν κατέστη δυνατό να συμφωνήσουμε σε όλες. Νομίζω ότι μπορεί να επιδειχθεί ρεαλισμός και από τις δύο πλευρές και θα πρέπει με επικοδομητικό τρόπο να σεβαστούμε τις κατευθυντήριες γραμμές μας και τις ε, κόκκινες γραμμές μας που έχουμε διαμορφώσει από το παρελθόν. Σεβόμεθα το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, αλλά θεωρούμε τον Brexit ένα ιστορικό λάθος, το οποίο δυστυχώς θα αντιμετωπίσει με αρνητικό τρόπο τον Βρετανικό λαό. Ε, το άρθρο 50 δεν μπορεί να αλλάξει έτσι όπως είναι τώρα και αν ε, δεν μπορούμε στη Βρετανική Βουλή να βρούνε μια λύση από εδώ και πέρα τότε ίσως θα πρέπει να υπάρξει δυνατότητα είτε νέων εκλογών είτε νέου δημοψηφίσματος. Η πολιτική μας ομάδα είναι ξεκάθαρη ότι αν μια διεύρυνση του άρθρου 50 είναι κάτι το οποίο απαιτείται έτσι ώστε να δοθεί χρόνος για τις δύο αυτές επιλογές, για οποιαδήποτε από τις δύο αυτές επιλογές, φυσικά θα συμφωνήσουμε. Αλλά μια παράταση θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένη και όχι για να χάσουμε ακόμα περισσότερο χρόνο. Το Brexit είναι σε αδιέξοδο. Τώρα ε, θα πρέπει το Ηνωμένο Βασίλειο να δείξει υπεύθυνη η ηγετική θέση, να ξεκαθαρίσει τις επιθυμίες της και να προσπαθήσει να οδηγήσει τη χώρα εκτός των δυσκολίων. Εμείς θα παραμείνουμε αξιόπιστοι εταίροι, θα παραμείνουμε επικοδομητικοί εταίροι, εργαζόμενοι υπέρ των συμφερόντων των ευρωπαϊκών λαών. Από πλευρά των Ευρωπαίων Συντηρητικών, ο κύριος Κάμαλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Τίμερμανς. Καταρχά να ευχαριστήσω και τον κύριο Μπαρνιέ και τον κύριο Τίμερμανς για τι μετρημένε ομιλίε του. Νομίζω ότι ήταν πολύ σωστοί και δεν νομίζω ότι μπορεί να διαμαρτυρηθεί κανεί ε, για αυτά που είπαν. Να σα ε, μιλήσω ω κάποιο που παρατήρησε τη συζήτηση για την συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου από τι δύο πλευρέ ε, τη μάχη, Έχω μιλήσει με πολλά άτομα και από τι δύο πλευρέ των διαπραγματεύσεων και προτείναμε λύσει για να ξεπεράσουμε κάποιε δυσκολίε Και ω επικεφαλή τη ομάδα μου δεν ε, σας είπα μόνο με τι είμαστε αντίθετοι, αλλά πρότεινα και εναλλακτικέ λύσεις. Από τότε που έγινε ευρωβουλευτής, κάτι που μου έκανε εντύπωση στις σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζεται από τις δύο πλευρές της μάχης. Πολλοί πιστεύουν στο μοντέλο ε, πολιτικής ενοποίηση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενώ στα τελευταία 40 χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο η πολιτική τάξη ε, παρουσιάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως χώρο εμπορίου. Δεν αναφέρονται ή υποτιμούν την πολιτική ενοποίηση. Το γεγονό ότι η πολιτική έχει να κάνει με το πώ αντιλαμβάνονται οι συμπολίτε, έχει να κάνει επίση με το πώ αντιμετωπίζεται από τι δύο πλευρέ η αποχώρηση. Από ε, αυτή την πλευρά είπε σαφώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλουν να τιμωρήσουν κανένα, αλλά όποιο ε, αποχωρεί δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται όπω αντιμετωπίζονται τα μέλη. Είχατε μια ε, σκληρή στάση διαπραγματεύσει. Όχι μόνο γιατί είναι καλό αυτό για οποιοδήποτε διαπραγματευτεί, αλλά ούτω ώστε οποιαδήποτε συμφωνία να είναι αντικίνητρο για οποιαδήποτε άλλη χώρα θα μπορούσε να σκεφτεί ότι θέλει να αποχωρήσει. Οι περισσότεροι εδώ στο Κοινοβούλιο χαίρονται που οι στόχοι αυτοί επετεύχθησαν. Αλλά μου τονίζουν ότι έγιναν και συμβιβασμοί στην πορεία. Ορισμένοι ανησυχούν ότι το Μπάκστοφ μπορεί να δώσει ε, ένα αθέμητο προτέρημα στις βρετανικές επιχειρήσεις που θα έχουν πρόσβαση στην ενιαία αγορά. Άλλοι θεωρούν ότι μπορεί να μειώσει τη δυνατότητα στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνάψει συμφωνίε και μου είπαν ότι ελπίζουν δεν θα χρειαστεί το backstop. Το είπαν πολλοί ομιλητέ εδώ. Αλλά στο Westminster οι αντίπαλοι αυτή ε, τη συμφωνία το βλέπουν πολύ διαφορετικά. Για άλλη μια φορά είναι πολύ μεγάλο το χάσμα στην, ε, στο πώ αντιλαμβάνονται οι δύο πλευρέ. Θεωρούν ότι είναι μια ε, συμφωνία αποχώρηση με νομικέ υποχρεώσει που θεωρούν ότι μπορούν να του εμπλέξει σε μια τελειωνιακή ένωση για πάντα. Ορισμένοι υπεύθυνοι τη Κομισιόν είπαν ότι η τελειωνιακή ένωση θα είναι η βάση για τη μελλοντική σχέση και θεωρούν ότι το κείμενο αυτή τη συμφωνίας δεν περιέχει την υποχρέωση να περάσουμε σύντομα σε ε, συμφωνία ελευθέρου εμπορίου. Λένε ότι ναι μεν οι ε, συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το άρθρο 50 για να φύγει κανείς ε, όταν θέλει, ενώ η συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο δεν δίνει καμία δυνατότητα αποχώρηση από τον backstop και θεωρούν ότι δεν σέβεται και τους πολίτες της Βόρειας Ιλανδίας που είναι υπέρ της Ένωσης τη συνέχιση της ένωσής τους με το Ηνωμένο Βασίλειο. Και θεωρούν και μου το λένε ότι δεν χρειάζεται καθόλου backstop. Εφόσον ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός είπε ότι δεν θα υπάρξουν σκληρά σύνορα εάν δεν υπάρξει αποχώρηση με συμφωνία. Πολλοί λοιπόν ε, στην Βρετανική Βουλή που πολλοί τους θεωρούν και οπαθής, ε, θεωρούν ότι η έλλειψη συμφωνίας είναι καλύτερη από μια κακή συμφωνία. Όμως είδαμε και ότι το εργατικό κόμμα αξιοποιεί οποιαδήποτε ευκαιρία για να δημιουργήσει δυσκολίες στην κυβέρνηση. Ήδη έκαναν προτάσεις μομφής και άλλοι πολιτικοί θεωρούν ότι το Κοινοβούλιο ναι μεν ψήφισε υπέρ του Brexit χωρίς να κατανοεί ποιες είναι οι επιπτώσεις του. Θεωρούν λοιπόν ότι μπορούν να αντιστρέψουν το αποτέλεσμα της ε, ε, του δημοψήφισματος αυτού. Είμαστε σε μια κρίσιμη φάση διαδικασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ε, πολύ υπομονητική. Αλλά θα χρειαστεί να περιμένετε λίγο περισσότερο. Πρώτα απ' όλα να δούμε τι θα γίνει με την ε, πρόταση εμπιστοσύνη που πιστεύω θα την κερδίσει. Και κατόπιν η Πρωθυπουργό θα κάνει συζητήσει με όλα τα άλλα πολιτικά κόμματα για να βρει συμφωνία. Άρα έχετε μια επιλογή. Μπορείτε να μην κάνετε τίποτα, να προετοιμαστείτε για την έλλειψη συμφωνία. Μπορείτε να θεωρήσετε ότι μπορεί να σταματήσει το Brexit ή να, να αντιμετωπίσετε μερικέ από τι ανησυχίε των Βρετανών. Για παράδειγμα, να εξηγήσετε στον Ηνωμένο Βασίλειο ότι δεν θέλετε να του κρατήσετε για πάντα στην Ελληνική Ένωση και το backstop θα είναι προσωρινό. Καταλαβαίνω ότι ε, μπορεί να σα φαίνεται ότι σα ζητάω πολλά, γιατί θεωρείτε ότι είναι καλή συμφωνία που προσφέρετε στον Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά όπω και το 2015, όπου εάν είχαν γίνει κάποιε μικροαλλαγέ στι ε, διαπραγματεύσει με τον David Cameron, μπορεί να είχαμε αλλάξει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματο, νομίζω ήταν πραγματικά κρίμα αν δεν κάνετε περαιτέρω προσπάθειε για να καταλήξουμε σε συμφωνία που θα βοηθήσει τη Βρετανίδα Πρωθυπουργό να φτιάξει, ε, να δημορφώσει πλειοψηφία στο Westminster. Θέλουμε κυρίω ε, αυτό που μα ενδιαφέρει να, είναι, να εστιάζουμε στου πολίτε. Οι αποφάσει μα τι επόμενε μέρε και εβδομάδε θα επηρεάσουν τι δουλειέ, τι επιχειρήσει, την ανάπτυξη τη οικονομία μα. Η επιστολή τη Δευτέρα από του Προέδρου Τούσκ ε, και Γιούγκερ ε, έκανε κάποιε νήξει για περαιτέρω ευελιξία. Α ελπίσουμε ότι αυτή η ευελιξία μπορεί να μεταφραστεί σε συγκεκριμένε προτάσει για να αντιμετωπίσουμε τις ε, ανησυχίε που οδήγησαν στο αποτέλεσμα τη χθεσινή ψηφοφορία. Μόνο τότε θα σταματήσουμε να κοιτάζουμε το παρελθόν και θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μια πιο ειλικρινή σχέση για το μέλλον. για τους Ευρωπαίους Φιλελεύθερους και Δημοκράτες ο κ. Φερχόστατ. Ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Είχαμε ελπίσει ένα άλλο αποτέλεσμα, αλλά ε, βλέπουμε τώρα ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα της ε, ψηφοφορίας και στην Μεγάλη ε, Βρετανία ε, δεν ε, είχε ήδη μια άποψη σχετικά με το αποτέλεσμα και το τι θα συνέβαινε. Θα πρέπει να σας πω ειλικρινά, δεν έχω εκπλαγεί διότι από το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος είδαμε τι ε, γίνεται στο Whitehall, τις επενδύσεις και είχαμε πάντοτε πλειοψηφίες εναντίον, εναντίον ε, της ιδιότητας ε, του μέλους ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Τελωνιακή Ένωση, στην ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων, το Ιρλανδικό backstop και ο κατάλογος είναι πολύ μακρύς. Στη συζήτηση σήμερα το πρωί, κύριε Καμάλ, το ερώτημα είναι πώς να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο και ήλπιζα ότι θα μας δίνατε μια ένδειξη στην παρέμβασή σας. Περιγράψατε την κατάσταση, παρακολουθούμε, αλλά πώς θα βγούμε από αυτό το αδιέξοδο, πώς θα αποφύγουμε το καταστροφικό no αυτό το σενάριο και νομίζω ότι η απάντησή μου και νομίζω ότι θα συμφωνείτε μαζί μου χρειαζόμαστε μια μεγάλη πλειοψηφία υπέρ κάποιου, κάποιας λύσης ε, στην Βουλή των Κοινοτήτων και στην Βρετανική πολιτική. Μια πλειοψηφία προς όφελος ε, της Ένωσης και της Βρετανίας μπορούν να επιτευχθούν εάν τα πολιτικά κόμματα, όλα τα πολιτικά κόμματα στη Βρετανία, όχι μόνο το συντηρητικό, αν τα πολιτικά κόμματα αρχίζουν να βάζουν τα συμφέροντα του λαού και της Βρετανίας υπεράνω των στενών κομματικών συμφερόντων. Ας ε, το πω διαφορετικά. Ο κύριος Τζέρεμι Κόμπεν θέλει να γίνει πρωθυπουργός αυτής της χώρας η κυρία Μέη ε, θέλει να παραμείνει. Ε, βεβαίως είναι νόμιμο, ομνόμιμα όλα αυτά αλλά μερικοί θέλουν ε, να χρησιμοποιήσουν αυτό για μια ανεξάρτητη σκοτία. Είναι νόμιμα ότι θέλει να διατηρηθεί η ενότητα της χώρας. Όλα αυτά είναι νόμιμα. Αυτές οι νόμιμες φιλοδοξίες που έχουν όλες είναι όλες νόμιμες. Αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι ότι το αποτέλεσμα τώρα ε, θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που να τα υπερβαίνει όλα αυτά. Ένα σύστημα ε, που ε, υπεράνω του συστήματος που παρήγει ανταγωνισμούς. Βεβαίως υπάρχει μια, ένας ανταγωνισμός στο συντηρητικό κόμμα ε, στην πλάτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην αρχή της συζήτηση. Σήμερα έχουμε κάτι διαφορετικό. Δεν πρόκειται για μια ε, μάχη μέσα στο κόμμα. Είναι πρόβλημα υπαρξιακό της Βρετανίας, του μέλλοντος της ε, Βρετανίας. Της, δεν, δεν πρόκειται πια για μια μάχη. Εγώ βεβαίως ένας ταπεινός Βέλγος δεν θα κάνω μάθημα στους Βρετανούς για το τι πρέπει να κάνουν, αλλά αλλά πιστεύω ότι ήρθε η στιγμή να πούμε στους Βρετανούς φίλους μας ότι για το καλό της Βρετανίας θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των κομμάτων στη Μεγάλη Βρετανία όπως το κάνουμε εδώ στο Κοινοβούλιο από την πρώτη μέρα. Να δούμε ποιες θα είναι οι σχέσεις ανάμεσα στους δύο. Να προσδιορίσουμε τις σχέσεις, να βρούμε τις κόκκινες γραμμές ε, που υπήρχαν από την αρχή Βεβαίω, νομίζω ότι σκληρή γραμμή είναι στο συντηρητικό σώμα και εμεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σα λέμε ότι είμαστε έτοιμοι ε, για μια βαθύτερη μελλοντική σχέση πιο βαθύτερη από ό,τι προβλέπεται. Μισελ στην ε, δήλωση ε, και που επιβεβαιώθηκε πριν λίγα λεπτά και αν υπάρχει στην Βουλή των Κοινοτήτων μια διακομματική πλειοψηφία για μια βαθύτερη τέτοια σχέση, είμαστε έτοιμοι να δεσμευθούμε για να συμβεί αυτό. Υπάρχουν ε, δύο μικρές ανησυχίες Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να υπάρξει ένα no deal. Είναι επίμαχο αυτό το θέμα ε, και για την ευρωπαϊκή πολιτική καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεστε περισσότερο χρόνο. Βεβαίως είναι κακή μέρα ε, να πάμε πέραν του άρθρου 50, ε, πέραν της ημέρας των ευρωεκλογών. Αυτό θα συνεχίσει την αβεβαιότητα για όλους τους επιχειρήσεις. Και δεύτερη ανησυχία είναι το συμφέρον των πελατών, των πελατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασίλου deal ή μη deal θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτω ώστε να διαφυλάξουμε τα δικαιώματα τους, τα δικαιώματα που υπάρχουν στη Συμφωνία Αποχώρησης. Με την Επιτροπή ΛΥΜΠ ε, θα ασχοληθούμε με το Βουλή των Κοινοτήτων, με την Επιτροπή τους για να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα, διότι νομίζω ότι όλοι οι πολίτες δεν θα πρέπει ποτέ, ποτέ να είναι τα θύματα των ε, πολιτικών και κομματικών ε, παιχνιδιών, όπως βλέπουμε σήμερα με τον Brexit. Ευχαριστώ πολύ. Για ε, την ομάδα των Πρασίνων, ο κύριος Λάμπερτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτό που είδαμε χτες ήταν ένα συνασπισμός απίθανος μελών του Βρετανικού Κοινοβουλίου που ψήφισαν μαζικά κατά ενός πράγματος. Αυτό το πράγμα είναι, αν θέλετε, μια ε, συμφωνία η οποία έλαβε, λάμβανε υπόψη τους περιορισμούς τους νομικούς ε, του Good Friday Agreement. Η κόκκινη γραμμή της Βρετανικής κυβέρνησης αυτή καθεαυτή. Είδαμε ότι ε, προσπαθούμε ε, να διαφυλάξουμε την ακεραιότητα και τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό οδηγεί σε τη μόνη δυνατή συμφωνία. Και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζουμε στεναρά αυτήν την συμφωνία ε, που παρουσίασε ο Μισελ. Δεύτερο σημείο. Βλέπω ότι μια τροπολογία που κατατέθηκε που ήταν για την δημιουργία μιας δυνατότητας για το Ηνωμένο Βασίλειο μονομερός να βγει από το Good Friday Agreement απορρίφθηκε. Αυτό με ενθαρρύνει. Βλέπω ότι από τις δύο πλευρές της μάχης υπάρχει αποφασιστικότητα να διαφυλαχθεί αυτή η συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής και μην υποτιμάται τις δυνατότητες που μια δράση μονομερής θα μπορούσε να οδηγήσει και στην Ιρλανδία σε ε, βία. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια μεγάλη πλειοψηφία υπέρ ενός no deal σενάριο. Ένα τέτοιο σενάριο είναι αυτό που αυτόματα ε, λόγω ελήψεως άλλου θα συμβεί αν δεν υπάρχει πλειοψηφία θετική για μια εναλλακτική λύση. Μια εναλλακτική λύση που θα απαιτήσει από τις αρχές της Μεγάλης Βρετανίας να αναθεωρήσουν τις προσδοκίες τους για μια μελλοντική σχέση. Αντιβουλή των Κοινοτήτων είναι είτε πρόθυμη ή ανίκανη να βρει μια τέτοια θετική πλειοψηφία τότε ως δημοκράτης πιστεύω ότι η μόνη εναλλακτική θα είναι τότε να ζητήσουμε από το Βρετανικό λαό να επιλέξει αν θέλει το Brexit σύμφωνα με τις γραμμές που διαπραγματεύτηκαν τόσο η Βρετανική κυβέρνηση ναι, έτσι καταλαβαίνω τις βρετανικές παραδόσεις ως φιλοφρόνηση και fair play. Ε, νομίζω ότι ε, είχα αρκετό μερίδιο ε, παρέμβασης των ομιλιών μου από τους βουλευτές τους Βρετανούς. Θα ήθελα να δείξουν προσήλωση στις παραδόσεις τους. Γι' αυτό θα ήθελα να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι μπορείτε να προσφέρετε πολλά στην Ένωσή μας. Νομίζω ότι θα πρέπει ίσως να αποφασίσει ο Βρετανικός λαός μεταξύ του Brexit έτσι όπως έχει ε, συμφωνηθεί ε, η νέα ε, επιλογή. Νομίζω δεν λέχθηκαν πολλά για την οικονομία, της επιχειρήσης. Θα ήθελα όλοι μας από τις δύο πλευρές της μάχης να λάβουν υπόψη τους 3 εκατομμύρια πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και 2 εκατομμύρια των Βρετανών που βρίσκονται από αυτή την πλευρά, διότι αυτοί είναι όμοιροι ε, με αυτή την κατάσταση και θα πρέπει αυτό να μας υπενθυμίσει ότι η δημοκρατία και η πολιτική πρέπει να να αναφέρεται κυρίως στην ευημερία και την ευζοία των πολιτών μας. Για την ενιαία Ευρωπαϊκή Αριστερά το λόγο έχει η κυρία Άντερσον. Υποστηρίζουμε εμείς τον backstop γιατί είναι ο λιγότερο βλαπτικός τρόπος για να συνεχίσουμε. Αλλά δεν πρέπει να αποδυναμωθεί, δεν πρέπει να γίνει νέα διαπραγμάτευση. Καθημερινά η Βρετανική κυβέρνηση περιφρονεί τον λαό της Ιρλανδίας και αγνοεί τις προβλέψεις της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής. Το τμήμα του Βρετανικού κατεστημένου, το οποίο υποστηρίζεται από τον DUP, πάντα ήταν εναντίον της συμφωνίας αυτήν. Κάποιοι θεωρούν ότι το Brexit είναι μια καλή ευκαιρία για να απαλλαγούν από τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Δεν υπήρξε ποτέ θετική λύση για την Ιρλανδία από τη Βρετανική Βουλή. Ποτέ στο παρελθόν και ποτέ δεν θα υπάρξει και στο μέλλον. Αυτά τα παιχνίδια, τα απαράδεκτα στο Westminster ε, συνεχίζονται ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να υποστηρίζει τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής και υπάρχει κάτι στη Συμφωνία αυτή που δίνει μια λύση, δίνει μια διέξοδο. Και κύριε Φερχώστατη είναι και νόμιμη και δημοκρατική. Λέγει ότι αυτή τη στιγμή ο Υπουργό Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου θεωρεί ότι έχουν υπάρξει αποδείξιμες αλλαγές σε επίπεδο νοοτροπιών και στάσεων θα προκαλέσει ένα δημοψήφισμα για την Ιρλανδική ενότητα. Έχει υπάρξει τέτοια απόδειξη αλλαγής το γνωρίζει η Τερέζα Μέη, το είπε δημόσια, το γνωρίζει η Κάριν Μπράντλεϊ. Η, η Ιρλανδική κυβέρνηση πρέπει να λάβει υπόψη περισσότερο τη δήλωση του Συμβουλίου του Απριλίου 17, το οποίο λέει ότι σε περίπτωση που υπάρξει μια επιτυχής ψηφοφορία επί της Ιρλανδικής Ενότητας, τότε ο, ο βορράς της Ιρλανδίας θα παραμείνει τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν τω μεταξύ η Ιρλανδία έχει ανάγκη από έκτακτα μέτρα έτσι ώστε να γίνει σεβαστή συμφωνία στο σύνολό της, η συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε και να στηρίξουμε τη διεξαγωγή ενός δημοψηφίσματος για την Ιρλανδική Ενότητα. Έχουμε λοιπόν το δικαίωμα να αποφασίζουμε για το μέλλον μας χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις. Αυτό το προβλέπει η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Να προσπαθήσουμε λοιπόν να καθορίσουμε την ένωση στην οποία θέλουμε να ανήκουμε. Ο James Κόνολι έχουν μεγαλύτερη σημασία κάθε μέρα. Είπε ότι η Βρετανική κυβέρνηση δεν έχει κανένα δικαίωμα στην Ιρλανδία. Δεν είχε κανένα δικαίωμα στην Ιρλανδία και δεν θα έχει ποτέ κανένα δικαίωμα στην Ιρλανδία. Per il gruppo e για την Ένωση για την Ελευθερία και την Άμεση Δημοκρατία, ο κύριος Φαράζ. Εξοχότατε κύριε Μπάγνιε, εξοχότατε κύριε Τίμερμαντς. Αυτή είναι η όρη που χρησιμοποίησε η Βρετανή η Πρωθυπουργό ε, στην επιστολή επαιτίας που έστειλε πριν ε, από μερικές μέρες. Αξιοποίησε αυτούς τους όρους και αυτό είναι απόλυτα συνεπές με όλη τη διαπραγμάτευση που έκανε. Κατάλαβα στις 8 Δεκεμβρίου του 2017 που θα πήγαινε αυτή η διαδικασία για να τηρήσουμε μια προθεσμία που είχε θέσει ο κύριος Μπαγνιέ ο οποίο είναι ένας μη εκλεγμένο καρδιοκράτη των Βρυξελών, η κυβέρνηση, ε, συγγνώμη, η Πρωθυπουργό, έφυγε στις 4 πατέρα το πρωί για να σας βρει και υπέγραψε την αρχή του Ιρλανδικού backstop. Είχε πουληθεί η κατάσταση από τότε. Από τότε δεν έχουμε καμία ηγεσία. Και ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι δεν έμαθε το ιστορικό λάθος, δεν έμαθε το ε, ιστορικό δίδαγμα ότι όταν υποκύπτεις αυτούς που σε απειλούν, τότε θα σε απειλήσουν ακόμη περισσότερο. Το κείμενο αυτό ήταν ένα κείμενο παράδοσης και το έσκησε χθε η Βουλή των Κοινοτήτων. Είναι σαφέ από ό,τι είπατε ότι δεν θα κάνετε περαιτέρω παραχωρήσει όπω αυτή περιμένει. Αλλά εξακολουθεί να είναι πρωθυπουργό μα. Και αυτό από μόνο του είναι αξιοσημείωτο. Αν είχε αίσθηση τιμή, θα είχε φύγει τουλάχιστον θα, θα έπρεπε να έχει φύγει μέχρι σήμερα το μεσημέρι. Ορισμένοι λένε ότι κύριε Μπαρνιέ, ε, μα στην ουσία σπαταλήσατε δύο χρόνια τη ζωή σα. Δεν ισχύει αυτό γιατί νομίζω ότι πραγματικά τα φέρατε τα πράγματα όπως θέλατε. Και παρά το ότι 500 ε, βουλευτές ψήφισαν υπέρ του άρθρου 50. Αυτό αποδεικνύει ότι θα πρέπει μετά από δύο χρόνια ή να έχουμε μία ε, συμφωνία ή απλώ να σηκωθούμε να φύγουμε. Και αυτό το λέει και η συμφωνία αποχώρηση του Βρετανικού Κοινοβουλίου που λέει ότι θα φύγουμε χωρί όρου στι 29 Μαρτίου. Αλλά βέβαια εσεί λέτε ότι δεν υπάρχει στήριξη για έλλειψη συμφωνία. Αλλά νομίζετε ότι δεν υπήρχε στήριξη για τον Brexit. Μπορεί να εκπλαγείτε για το πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η κοινή γνώμη. Κύριε Τίμερμαντ, λέτε ότι αυτό θα κάνει μεγάλη ζημιά αλλά αν ε, όπω ε, είναι νομική μα υποχρέωση αποχωρήσουμε χωρί συμφωνία, θα γίνουμε μια ανεξάρτητη χώρα. Δεν έχει τιμή, δεν έχει τίμημα η ελευθερία. Αλλά παραδέχομαι ότι αμφιβάλλουν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Γιατί βεβαίω ε, στην ουσία τα έχουν βρει μαζί σα. Είναι επίση και ο κύριο Μπλεαρ και πολλοί άλλοι από το Βρετανικό κατεστημένο που θεωρούν ότι η ψήφο για τον Brexit και γενικά η εκλογή είναι αξιοπεριφρόνητη. Και υπάρχει θαυμάσια παράδοση. Το είδαμε με τη Δανία, το είδαμε με την Ιρλανδία. Του βάζετε να ξαναψηφίσουν. Τι μπορώ να πω. Αν τελικά καταλήξουμε με παράταση του άρθρου 50, μπορεί να καταλήξουμε να συμμετάσχουμε και στι επόμενε ευρωεκλογέ. Και θα συμμετάσχουμε. Και αν η προδοσία γίνει τέλεια και αν χρειάζεται να κάνουμε δεύτερο δημοψήφισμα, τότε μπορεί να αντιμετωπίσετε μια μεγάλη έκπληξη. Μπορεί να είναι πολύ ήρεμοι και χαλαροί οι Βρετανοί, αλλά άμα τους πιέσει, τότε γίνονται λιοντάροι που θα χυμίξει να σας φάει. Θα γίνουν ακόμη πιο ανεξάρτητοι αν γίνει δεύτερο δημοψήφισμα και θα το κερδίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη πλειοψηφία. για την ε, ε, ομάδα της Ευρώπης των Εθνών. Για την ομάδα της ε, Ευρώπης των Εθνών και της Ελευθερίας, ο κύριος Μπάτεν. Ευχαριστώ. Half years of an elaborate political charade. Εδώ για δυόμιση χρόνια έχουμε καραγκιοζουλίκια. Με βάση λάθο προποθέσει. Ότι δεν μπορεί να φύγει κανεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρί συμφωνία. Μα δεν πρόκειται ποτέ να προκύψει συμφωνία. Δεν θα προκύψει συμφωνία. Η κυρία Μέη και οι διάφοροι απεσταλμένοι του πηγαίνουν προ πίσω, Βρυξέλλε, Λονδίνο, για να καταλήξουν σε μια συμφωνία από χώρε που κανεί δεν τη θέλει. Δεν τη θέλουν αυτοί που θέλουν να παραμείνει, εφόσον δεν θέλουν να φύγει. Δεν τη θέλουν αυτοί που θέλουν να φύγουν, γιατί στην ουσία έτσι δεν φεύγουμε με τέτοια συμφωνία. Και τι εξυπηρετούν όλα αυτά. Θα γίνει παράταση. Ούτω ώστε τελικά ε, μέσω φθορά ε, να ε, αντιστρέψετε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματο. Να κουράσετε του εκλογεί. εκλογείς. Για πρώτη φορά συμφωνώ με κάτι που λέει ο κ. Φερχόφστατ. Πώ να ξεπεράσουμε το αδιέξοδο. Στο Βρετανικό Κοινοβούλιο χρειαζόμαστε μια πλειοψηφία υπέρ κάποιου πράγματο. Απόλυτα σωστό κύριε Φερχόφστατ. Σε τρει μέρε η κυρία Μέη πρέπει να μας υποβάλει ένα δεύτερο σχέδιο, ένα plan B. Υπάρχει ένα plan B που θα έπρεπε να είναι το plan A. Θα ήταν να καταργήσουμε το νόμο του 1972 για τη συμμετοχή στην Ένωση και τότε θα αποχωρήσουμε με βάση τους δικούς μας όρους και μετά θα δούμε πώς θα καταργήσουμε, θα τροποποιήσουμε με βάση τις δικές μας προτεραιότητες τις δεκάδες χιλιάδες νομοθετήματα που έχουμε υιοθετήσει έκτοτε με το δικό μας χρονοδιάγραμμα. Θα πρέπει να παραιτηθεί αμέσως η κυρία Μέη και να γίνει πρωθυπουργός κάποιος που να θέλει να φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Βρετανικό Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα να αποκαταστήσει την τιμή του. Αν προδώσει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, θα καταστρέψει οποιαδήποτε αξιοπιστία υπάρχει ακόμη για το δημοκρατικό μα σύστημα, που δεν είναι και πολύ υψηλή, αλλά μπορούν να αντιστρέψουν την κατάσταση, μπορούν να πάρουν την πρωτοβουλία, μπορούν να σταματήσουν να σα ζητάνε να του πείτε πώ θα φύγουμε και να αρχίσουμε να λέμε εμεί πώ θα φύγουμε. Και ο λαό μα ποτέ δεν θα παραδοθεί. Η κυρία Ντότς, μία εγγεγραμμένη. Ευχαριστώ όσους από την, την Επιτροπή και το Συμβούλιο για τη συνεισφορά τους. Ε, το βράδυ έχουν απορρίψει την ε, συμφωνία. Κάνοντας το αυτό, υποστήριξαν την ακαιρεότητα, την ε, συνταγματική θέση της Βόρειας Ιρλανδίας, ε, την ενότητα της ενιαίας αγοράς της Βρετανίας και την προσδοκία για ένα ανεξάρτητο μέλλον εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα το πρωί υπάρχει κάποια σύγχυση σχετικά με την νομική θέση της, της Ηνωμένου Βασιλείου, σχετικά με την παράταση του άρθρου 50 νέου δημοψηφίσματος. Είναι η νομική θέση που θα, από την οποία θα φύγει στις 29 ε, Μαρτίου το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι σαφές στοιχείο ε, του νόμου. Δεν πρέπει να υπάρχει σύγχυση. Υπάρχει επίσης η πρόταση backstop. Έγινε πολύ λόγος ε, για ε, βία εάν δεν επιτύχει αυτό που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς στο DUP δεν θέλουμε σκληρά σύνορα. Και νομίζω ζητώντας το backstop δεν υπάρχει επιλογή no deal επιτάπητος μην ε, επιτρέποντας ε, βιώσιμες αλλαγές, νομίζω έγινε αναπόφευκτο το αποτέλεσμα της χθεσινής ψηφοφορίας. Όλες οι πλευρές είπαν ότι δεν πρέπει να υπάρχουν σκληρά ε, σύνορα με οποιοδήποτε σενάριο. Δεν θα πρέπει να προσπαθούμε να ελαχιστοποιούμε όλες τις τριβές στα σύνορα χωρίς ε, το επίμαχο θέμα του backstop. Νομίζω αυτή ήταν η απάντηση πάντοτε ε, και έτσι ε, θα μπορέσουμε να έχουμε πρόοδο. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Έλμαρ Μπρόκ. Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, αγαπητέ Μισολμπάνια, συνάδελφοι. Νομίζουμε ότι από τη συζήτηση καθίσταται σαφές, όπως και από πολλές πρωτεύουσε, ότι υπάρχει ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 27 κράτη-μέλη έχουν την ίδια αντίληψη. Αλλά στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπάρχει ενότητα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εμείς θα εμείνουμε στην ενότητά μας και στην ε, ε, ακαιρεότητα της ε, ενιαίας αγοράς. Το δεύτερο. Χθες Υπήρξε μια συμμαχία ε, των αρνητών. Από τη μία είναι οι σκληροί αποχωρητές, από την άλλη είναι αυτοί που θέλουν να παραμείνουν και συμφωνούν σε αυτό που δεν θέλουν. Η Τερίζα Μέη προσπάθησε να προσφέρει μια ε, επικοδομητική λύση. Τώρα όμως λέει ότι θα μιλήσει με την αντιπολίτευση. Θα πρέπει να έχει μιλήσει από δύο χρόνια. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια οικονομική λύση από το Βρετανικό Κοινοβούλιο τελικά επί της οποίας να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Ο κύριος Κόρμπιν είπε ότι θέλει η Τελωνιακή Ένωση. Ε, κάνει αυτή την πρόταση. Ας βρει πλειοψηφία για αυτήν. Δεν θα είχαμε πρόβλημα. Και θα μας επέτρεπε να βρούμε μια λύση. Θα ήταν πολύ καλοδεχούμενο κάτι τέτοιο. Αν υπάρξει μια επικοδομητική λύση, βεβαίω να την εγκρίνουμε. Πέρασε τώρα η εποχή που θα έπρεπε οι κομματικές και προσωπικές φιλοδοξίες να αποτρέπουν την εξέβρεση λύσης. Πρέπει λοιπόν να τολμήσουν οι Βρετανοί να έχουν αυτό το θάρρος. Ο κύριος Βάιντενχολτσερ. Ευχαριστώ. Είναι ιστορική στιγμή. Όπως ξέρουμε η ιστορία πάντα μας εκπλήσει. Όταν ξεκινήσαμε τη θητεία μας το 2015, κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει ότι θα κάναμε σήμερα μια τέτοια συζήτηση. Ούτε καν το 2016, όταν συζητούσαμε το απροσδόκητο αποτέλεσμα του Βρετανικού Δημοψηφίσματος. Πέρασαν έκτοτε 900 μέρες μέχρι να λάβει μια απόφαση που να έχει έννοια το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Περάσαμε μήνες αβεβαιότητας και το αποτέλεσμα είναι σαφέ το μέλλον εξακολουθεί να είναι απρόβλεπτο. Απόλυτα σκοτεινό. Ένα όμως είναι σαφές. Τελειώνει ο χρόνος. Θα λήξει ο χρόνος. Σε 70 μέρες υπάρχει κίνδυνος να υπνοβατήσει αυτό το μεγάλο έθνος προς την καταστροφή. Θα πρέπει να καταλάβετε ως καμπανάκι αυτά που έγιναν χθε. Θα πρέπει να συζητήσουμε τη λογοδοσία ε, των κυβερνητών. Πώς είναι δυνατόν μια μικρή ελίτ για κοντόθωρους λόγους να έχει όμοιρο ολόκληρη τη χώρα. Είναι σαφές ότι απέτυχαν οι Βρετανοί συντηρητικοί. Αλλά τώρα το θέμα δεν είναι να επιμένουμε ποιος έχει δίκιο, ούτε να επιχειρήσει κανείς να εκδικηθεί ή να επιβάλλει αντίπεινα. Πρέπει να δράσουμε υπεύθυνα προς το συμφέρον των πολλών και όχι των λίγων. Οι απλοί άνθρωποι στη Βρετανία έχουν πολλά να χάσουν εάν υπάρξει σκληρή αποχώρηση. Εμείς, τα 27 κράτη-μέλη που μείναμε ενωμένοι καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων πρέπει να είμαστε ευέλικτοι για να ξεπεράσουμε το αδιέξοδο και για να υπάρξουν πραγματιστικέ λύσει να ελαχιστοποιήσουμε τι ζημίες. μπορείτε να βασιστείτε στην ομάδα τη δική μα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Τα τελευταία 40 χρόνια δεν ξεχνάμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει συμβάλει τρομερά στο κοινό μα εγχείρημα. Θα μα λείψει η εμπειρογνωμοσύνη των Βρετανών συναδέλφων μα, Αλλά η ζωή συνεχίζεται. Πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε αποτελέσματα στην προσπάθειά μα. Θέλουμε λοιπόν βεβαιότητα για το τι θέλει το Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλουμε σαφή μηνύματα. Θα μπορούσε μια νέα ψηφοφορία να μα δώσει αυτό το αποτέλεσμα, ένα νέο ψήφισμα. Ο, ο Βρετανικό λαό θα έπαιρνε την κατάσταση στα χέρια του και κανεί δεν θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι ε, δεν ξέρει γιατί ψηφίζει ο ψηφοφόρο. Δεν θέλω να παρέμβω στα εσωτερικά σας, αλλά θα καλοδεχόμεθα οποιαδήποτε απόφαση να παραμείνετε. Στείλαμε μία επιστολή μαζί με 40 συναδέλφους αυτή την εβδομάδα για να καταστεί σαφές ότι θέλουμε να μείνετε και θα σας καλωσορίσουμε με ανοιχτές αγκάλες εάν επανέλθετε. Κύριε Βάδεν Χόλτσερ, υπάρχει μια μπλε κάρτα. Θέλετε να απαντήσετε. Όχι, ευχαριστώ. Σας κατανοώ. Έχετε όλοι να αντιμετωπίσετε αυτές τις αχλαμάρες. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Αλλά παρατηρήσατε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι και τόσο ενωμένο και με την συντηρητική κυβέρνηση δυστυχώς έχει διαιρεθεί ε, ακόμα περισσότερο. Και εγώ εκπροσωπώ τη σκοτία ε, και η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Εμείς θέλουμε να μείνουμε στην Ηνωμένη Ευρώπη, θέλουμε να μείνουμε στην οικογένεια των ευρωπαϊκών κρατών. Αλλά έχετε να αντιμετωπίσετε το Ηνωμένο Βασίλειο ως έχει πρέπει να σεβαστείτε τη συνταγματική τάξη της συγκεκριμένη χώρας. Η θέση της Σκοτίας είναι σαφής. Δεν υπάρχει καλό Brexit. Είναι κακό για τη Σκοτία, κακό για το Ηνωμένο Βασίλειο, κακό για την Ενωμένη Ευρώπη. Η προσπάθειά μου δεν είναι να μετριάσω τις αρνητικές συνέπειες του Brexit, αλλά να σταματήσω τον Brexit. Και υπάρχουν πολλοί Βρετανοί οι οποίοι ανήκουν σε πολλά κόμματα συνάδελφοι που προσπαθούν να βρουν κάποια λογική λύση. Πρώτον, χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Λυπάμαι γι' αυτό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Άμα θέλετε να παραμείνουμε, θέλουμε χρόνο. Και ίσως να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τη διαδικασία αυτή μόνο αν συνεργαστούμε στενά και τότε ίσως η κυβέρνηση της, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου ακούσει και άλλες φωνές και όχι μόνο τις δικές της. Πάρα πολλοί πολίτες στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Υπήρου αγχώνονται οι Βρετανοί πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολίτες της Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε ευθύνε για την προστασία των δικαιωμάτων τους. Πρέπει να σεβαστούμε τα δικαιώματα αυτά, να διευκρινίσουμε την κατάστασή τους, να τους διασφαλίσουμε το μέλλον τους ε, και να μην τους δώσουμε την δυνατότητα να παραμείνουν μέσα σε μια διαδικασία την οποία δεν ελέγχουν. Είναι καθήκον προς τους πολίτες μας. Η Επιτροπή έκανε προσπάθειες για να υπάρξει εγγύηση για τα δικαιώματα αυτά, αλλά λόγω της απουσίας δράσης από πλευρά της Βετανικής κυβέρνησης πρέπει εμείς να αναλάβουμε δράση. Νομίζω ότι αυτά τα δύο, ε, οι δύο στόχοι αυτοί μπορεί ε, να βοηθήσουν. Θα πρέπει έτσι να βοηθήσουμε και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που δημιουργεί το Westminster. Έχετε μία μπλε κάρτα, θέλετε να απαντήσετε. Από ποιον είναι η μπλε κάρτα, λέει ο κ. Σμιτ. Όχι, όχι, δεν θα δώσω περισσότερο οξυγόνο στον Κόμπερν από όσον ήδη καταναλώνει. Η κυρία Σπινέλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η προοπτική μιας έλλειψης συμφωνία για τον Brexit αντιπροσωπεύει ένα, μια σοβαρή βλάβη για τη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής πάνω στην οποία οι κάτοικοι της Βόρειας Ιρλανδίας κάποτε θα κληθούν να αποφασίσουν, αλλά και για τους Βρετανούς πολίτες που ζουν ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ορίζοντας είναι σκοτεινός. Η απουσία μιας συμφωνίας θα του στερήσει τα δικαιώματα ελευθερίας διακίνησης. Από τη σημερινή εκκρεμότητα θα περάσουν στη νομική αβεβαιότητα, σε ένα εφιάλτη. Είναι δύσκολο να δούμε πώς θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την τεράστια σύγχυση την οποία έχει δημιουργήσει η εκτελεστική εξουσία αν δεν εκφραστεί για μια ακόμη φορά ο λαός. Αν επιβεβαιωθεί το no deal, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να προστατεύσουν τα δικαιώματα των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου ζητώντας να ευθυγραμμιστούν οι εθνικές πρακτικές στα λεγόμενα best practice και δίδοντας εγγυήσει στους Βρετανούς πολίτες για την ελεύθερη διακίνησή τους. Ακόμα πιο σοβαρή είναι η θέση των τριών εκατομμυρίων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο που κινδυνεύουν να βρεθούν και αυτοί θύματα του εχθρικού περιβάλλοντος που προωθούν οι συντηρητικοί από το 2012. Οι υποσχέσεις της ΜΕΙ μπορεί να αναιρεθούν με μια σύντομη ψηφοφορία από το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Μόνο αν εφαρμοστούν οι προβλέψεις της συμφωνίας θα τους δώσει μια νομική ασφάλεια. Η προστασία νομική των δικαιωμάτων αυτών είναι δυνατή εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύσει μονομερός τους πολίτες της Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρώπη και οδηγηθούμε εκ νέου σε μια προκαταρκτική συμφωνία Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου που προστατεύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το κεφάλαιο για τα δικαιώματα. Αυτό είναι κρίσιμο, αυτό είναι σημαντικό και γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε περισσότερο χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλω να ευχαριστήσω εδώ και το επαναλαμβάνω αυτό στον κύριο Μπαρνιέ. Η κυρία Άτκινσον έχει το λόγο. Δεν είμαστε λίγο ε, απογοητευμένοι σήμερα. Κυρία Μέη, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ιούνκερ, τον κύριο ε, Φερχόφσταντ, ε, οι οποίοι ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, του όσοι ψήφισαν 17 εκατομμύρια οι οποίοι ψήφισαν για το Brexit και να σας υπενθυμίσω ότι είμαστε GPOC, δεν είμαστε θηγατρικοί των κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπήρξε προδοσία. Έχουμε έχουμε μια κυβέρνηση, μια πρωθυπουργό και αντιπολίτευση 17,2 εκατομμύρια που ε, ψήφισαν ε, ή ψήφισαν μαζί με με, τους, αυτούς των Ηνωμένων Πολιτειών του Commonwealth. Μπορούμε ε, να ακολουθήσουμε τους κανόνες του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορία έχουμε του 17,4 εκατομμύρια που ψήφισαν για το Brexit. Θα κάνουμε και πάλι τη Μεγάλη Βρετανία μεγάλη. Θα ήθελα να ξαναγίνει μεγάλη η Μεγάλη Βρετανία και πάλι στον μεγάλο ευρύτερο κόσμο. Επόμενος ομιλητής για δύο λεπτά, ε, η κυρία Κέλλη. Ναι, ε, συμφωνώ με τα περισσότερα πράγματα που λέχθηκαν εδώ σήμερα. Θα ήθελα να πω ότι η ψηφοφορία εχθές το βράδυ ήταν κάτι το προβλέψιμο. Και οφείλω να ομολογήσω ότι η ενότητα των 27 είναι θαυμαστή χάρη στο Μισελ Μπαρνιέ, ε, στην εργασία του και στην εργασία όσων συμμετείχαν σε αυτό το έργο. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω. Θα ήθελα να επανέλθω σε ένα σχόλιο που λέχθηκε ε, χτες. Το να προσπαθήσει να πει κανείς αυτό σε αυτούς που ε, έχουν αυτά τα σύνορα που προστατεύονται από τους Βρετανούς ε, στρατιώτες το να πει κανείς ότι αυτά όλα δεν είναι χρήσιμα και χάρη σε βία που υπήρξε είχαμε τη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής και να πούμε ότι ο, ο κύριος Μπαρνιέ και ε, το, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, κάνανε το παν για να εξασφαλίσουν ότι θα προστατευτεί η συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής και η ειρήνη σε όλη την Ιρλανδία θα ήθελα να πω στην συνάδελφο Άντερσον ότι δεν είναι η στιγμή ε, να ε, κάνουμε τέτοια έκκληση. Δεν είναι η θέση ε, της Ιρλανδικής κυβέρνησης του λαού της Ιρλανδίας παρόλο που ευχόμαστε μια ενωμένη Ιρλανδία. Δεν νομίζω ότι αυτό ήθελε ο πληθυσμός. Ο μεγάλος φόβος είναι να μην υπάρξει συμφωνία το να βγει με τρόπο άτακτο από το Ευρωπαϊκή Ένωση η Μεγάλη Βρετανία. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο αποτέλεσμα. Αλλά ο φόβος είναι η Μεγάλη Βρετανία να λάβει μια απόφαση που δεν είναι πράγματι αυτό ε, που θέλει, αυτό που θέλει ο λαός. Δεν θέλει ένα τέτοιο σενάριο. Θα πρέπει να μπορεί να εκφραστεί και θα πρέπει ότι το πιο ε, έξυπνο θα ήταν να ξανασυμβουλευτούμε αυτούς που ψηφίσαν ο Βρετανικός λαός. Είναι πραγματικά αυτό που ήθελε, νομίζω ότι θα πει όχι αν ξαναερωτηθεί. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά στον κύριο Ντάντς. Ευχαριστώ. Ας είμαστε σαφείς. Πώς καταλήξαμε εδώ. Ε, η κυβέρνηση ενδιαφερόταν μόνο για τα συμφέροντα του Συντηρητικού Κόμματο και δεν τα προστάτευσε ούτε καν πολύ καλά. Έτσι καταλήξαμε εδώ. Η κυβέρνηση αυτή αρκεί, θα έπρεπε να φύγει. Αλλά αυτή η συζήτηση φυσικά πρέπει να γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οποιοδήποτε κόμμα είναι στην εξουσία θα πρέπει να κάνει αυτή την επιλογή σε σχέση με τον Brexit. Ή θα αποχωρήσει κανείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση καταστρέφοντας ε, θέσεις εργασίας, καταστρέφοντας το περιβάλλον, καταστρέφοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων ή παραμένεις εντός της Ένωσης και χάνεις οποιαδήποτε δυνατότητα να επηρεάσει αυτές τις δομές. Αυτή είναι η επιλογή εάν υπάρξει Brexit. Κανένα από αυτά τα δύο δεν είναι σωστά για καμία χώρα και σίγουρα όχι για το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά εγώ θέλω να σα δώσω ένα μήνυμα ελπίδα για την Βρετανία. Χάρη σε αυτού του τύπου απέναντι που είναι τόσο περίεργοι, καταλήξαμε στο μεγαλύτερο φιλοευρωπαϊκό κίνημα στην Ήπειρο. Έχουμε εκατομμύρια πολιτών μα που είναι δεδεθμένοι να βγουν έξω για να υπερασπιστούν τι αξίε τη Ένωση και να πούνε ανοιχτά ότι είμαστε περήφανοι για αυτά που έχει επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά που θα επιτύχει. Θα υπερασπιστούμε την ελεύθερη κυκλοφορία. Θα υπερασπιστούμε τι δομέ τη Ένωση, Όχι αυτέ που έχουμε τώρα, αλλά και αυτές που θα αποκτήσει το μέλλον η Ένωση. Και αυτές οι ανοησίες και ε, τα ψέματα που λένε, την άλλη μεριά, καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει πλειοψηφία για άτακτη αποχώρηση. Εάν θα υπάρξουν νέε εκλογέ, εάν θα υπάρξει νέο δημοψήφισμα, εάν θα υπάρξει νέα πλειοψηφία για κάποια άλλη λύση, χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Σα παρακαλούμε, συνάδελφοι, α μην αφήσετε τη διαδικασία να νικήσει την πολιτική. Έχουμε δυνατότητα να αντιστρέψουμε αυτή την πορεία. Θέλουμε τη στήριξή σα και τη φιλία σα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Σκοτ Κέιτσο, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είδα την ιστορική ψηφοφορία στο Westminster, εδώ στο Στρασβούργο με συναδέλφου ε, από όλε τι χώρε που ανησυχούν ιδιαίτερα για την κρίση αυτή. Πολλοί ελπίζουν να βρούμε έναν τρόπο να μείνουμε. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω για τη στήριξή σα. Το Brexit είναι η ε, αποτυχία τη ηγεσία. Απέτυχε η Τερίσα Μέη ασχολήθηκε μόνο με τις ανάγκες του κόμματός της. Ο Τζέρεμι Κόρμπιν απέτυχε στο συνταγματικό δικαίωμά του, ε, συνταγματική υποχρέωσή του να αντισταθεί στο Brexit. Η χώρα μας λοιπόν είναι σε απόγνωση, αλλά το Brexit είναι και έλλειψη αλληλεγγύης. Οι παλαιότερες γενιές αγνοούν τους πόθους των νέων. Πολλοί Βρετανοί ξέχασαν τους άλλους πολίτες που είναι στην κοινότητά μας και παίζουν ζωτικό ρόλο, ό, τους συναδέλφους, ε, τους συμπρατριώτες τους που ζουν εκτός ε, Βρετανίας. Πολλοί είδαν τη ζωή τους να αντιστρέφεται. Και τώρα που η περιπλοκότητα και το κόστος του Brexit κατέστησαν σαφή, πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε για τη χώρα μας. Είναι ε, απόλυτα απολωμένο και σε αδιέξοδο το Westminster. Πρέπει ο λόγος να επανέλθει στο Βρετανικό λαό. Ευχαριστώ πολύ. Δύο λεπτά, Γκονθάλεφ Πόντς. Αγαπητοί συνάδελφοι, χθε ε, είχαμε αυτή την ψηφοφορία που κατέστησε μόνο ένα σαφέ. ότι η Βουλή των Κοινοτήτων απέρριψε τη συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση, αλλά δεν ξέρει τι θέλει. Είχαμε πλειοψηφίε σε δύο αρνητικέ πλειοψηφίε, αλλά καμία πλειοψηφία για τη θετική ψήφο. Μετά από μήνε ε, αυταπατών και ψευδεστήσεων, θα πρέπει επιτέλου το Βρετανικό Κοινοβούλιο να αποδειχθεί την αλήθεια. Το Brexit δεν είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Είναι βρετανικό πρόβλημα. Οπότε σας παρακαλώ βρείτε λύση. Όλοι θέλουν ε, την καλύτερη δυνατή σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Όλοι το θέλουμε. Αλλά όχι πάση θυσία. Είμαστε φίλοι και σύμμαχοι. Αλλά αυτό που δεν μπορεί να αναμένει από εμά το Ηνωμένο Βασίλειο είναι να ε, καταρρύψουμε τις αρχές μας. Για έναν απλό λόγο. Το να είναι κανεί μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι οικονομική λύση. Είναι μια επιλογή ζωή. Είμαστε μια κοινότητα κοινών αξιών που βασίζονται στο κράτο δικαίου και συνθήκε. Δεν είναι απλώς εμπορική σχέση. Η Βρετανική κυβέρνηση δημιούργησε αυτό το πρόβλημα. Η Βρετανική κυβέρνηση πρέπει να το λύσει. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε τεθειμένοι να υπογράψουμε οποιαδήποτε συμφωνία αν έλθει σε εμά. Αλλά είμαστε και διατεθειμένοι να συνεχίσουμε χωρί συμφωνία. Μέχρι χθε θεωρούσαμε ότι το Brexit ήταν αντίδραση σε μια ευρωπαϊκή κρίση. Τώρα ξέρουμε ότι είναι αντίδραση σε μια εθνική βρετανική κρίση. Χθε κατέστη Αφές, ότι δεν υπάρχει πλειοψηφία για Brexit με συμφωνία και δεν υπάρχει συμφωνία για Brexit χωρί συμφωνία. Άρα το πιο λογικό θα ήταν να ηρεμήσετε και να συνεχίσετε να προσπαθείτε. Και στον κύριο Φαράτζ, δεν είναι εδώ βέβαια, με κάθε σεβασμό, σας παρακαλώ να είστε πολύ προσεκτικό όταν χρησιμοποιείτε τη λέξη πόλεμος. Γιατί ναι, υπήρξε πόλεμο. Και δόξα τω Θεώ, τον κέρδισαν οι Βρετανοί. Όλοι πήραμε το ε, μάθημα, αλλά ίσως όχι ο κύριος Φαράτζ. Κύριε Κονθάλεφ Πόντς, έχετε μια μπλε κάρτα. Από τον κύριο Έθεριτζ. Θέλετε να απαντήσετε. Φυσικά όχι. Είπατε όχι. Ω, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Θα πάω στον Οριλά. Ο κύριος Γκονθάλεφ Πόνς ε, είπε όχι. Ευχαριστώ. Και τώρα... Φεύγετε κύριε Έθελιντς. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, για δύο λεπτά, η κυρία Ντελάνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να πω ότι αυτό που συνέβη χτες στο, ε, στη Βουλή των ε, Κοινοτήτων ήταν κάτι το ιστορικό, κάτι που το περιμέναμε. Βεβαίως, συλλογικά δεν ξέρουν ε, τι θέλουν, μόνο ξέρουν να βγάζουν μεγάλους λόγους. Κάπως όπως ο κύριος Φαράζ, ο οποίος ακόμα και σε αυτή τη συζήτηση μια μισή ώρα για το Brexit. Το Brexit είναι raison d'être, δεν μπορεί να παραμείνει ε, σε αυτήν την αίθουσα. Ε, νομίζω ε, μας μίλησε, ήταν στο YouTube και έφυγε. Δεν ξέρει ο κύριος Φαράζ τι θέλει. Αυτό που θέλει είναι το πιο σκληρό Brexit με χωρίς συμφωνία, no deal, για να ε, μπορέσει ε, να καταστρέψει τις δουλειές ε, των συνειδητών ανθρώπων και να δημιουργήσει κάτι άλλο. Ακούγοντας τη συζήτηση εδώ σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτό που ακούω από τους συναδέλφους είναι Α καθίσουμε και ας δούμε τι μπορούμε να ε, συμφωνήσουμε για να υπάρξει μια πλειοψηφία και μια λύση. Ε, κάποιος λέει θα προτιμούσε μια τελωνιακή ένωση. Γιατί κανείς δεν προτείνει στη Βουλή των Κοινοτήτων μια τροπολογία γι' αυτό και να δει μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Μια τελωνιακή ένωση θα ήταν η καλύτερη ένωση να αποχωρήσουν οι Βρετανοί για να κρατήσουμε τις θέσεις εργασίας από τις δύο πλευρές της μάχης και να βρεθεί μια λύση. Ε, ασχολούμαστε ε, με πολιτική εδώ και στο Westminster όχι μόνο για να βγάζουμε λόγους αλλά για να δημιουργούμε πλειοψηφίες και να βρίσκουμε λύσεις. Ας αρχίσουμε να εργαζόμαστε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, περνάμε στη διαδικασία προσέγγιση του Προέδρου. Αν αυτό το χρόνο, θα ε, μιλήσω στον περισσότερο. Κύριο of Political... Οι Βρετανοί φίλοι μας βρίσκονται σε κατάσταση πολιτικής σύγχυσης σε σχέση με τον Brexit. Θα πρέπει να ανταποκριθούμε με δημιουργικό τρόπο. Πρώτον θα πρέπει να, προσθέσουμε, να δώσουμε στους Βρετανούς περισσότερο χρόνο για να αποφασίσουν. Δεύτερον, που αποφασίσουν κατά ε, του σκληρού Brexit, τότε θα πρέπει να συνεχίσουν να συμμετέχουν και στην ενιαία αγορά ε, και στην Τελωνιακή Ένωση φυσικά. Να δείξουμε ποια ήταν τα σοβαρά λάθη που έγιναν μέχρι τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πραγματικά ανάγκη το Ηνωμένο Βασίλειο και κάθε μέρα μας δείχνει ότι και το Ηνωμένο Βασίλειο χρειάζεται επίσης την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Λόπες Αγουιλάρα. Πρόεδρε, μια αρνητική πλειοψηφία από ετερόκλητους βουλευτές στην ουσία οδήγησε το Ηνωμένο Βασίλειο σε μια μακρά και σκοτεινή σύραγγα σύγχυσης και δημιουργούνται προβλήματα σε επίπεδο πολιτικό, σε επίπεδο κοινωνικό, σε επίπεδο οικονομικό και σε επίπεδο γενεών θα έλεγα και διαφορών μεταξύ τους. Η Βρετανική κυβέρνηση οδήγησε σε ένα δημοψήφισμα το οποίο δυστυχώς δεν έδωσε αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα. Υπάρχουν εκατομμύρια Βρετανών οι οποίοι άκουσαν με πάρα πολύ υπομονή τα ψέματα και τις ύποπτες δηλώσεις των εθνικιστών και των λαϊκιστών. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε ένα μήνυμα σαφές κατανοητό το οποίο να παρέχει ασφάλεια και εγγυήσεις. Πρέπει να σεβαστούμε τους πολίτες και να τους ελαφρύνουμε από τις επιπτώσεις της ανασφάλειας και της, του φόβου. Κύριος Γιούρεκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κρίση της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας είναι κάτι το οποίο διαπιστώνουμε εδώ. Μιλάμε για τον πλουραλισμό και τον διάλογο και κάθε φορά οι συνάδελφοι που ζητούν τον λόγο τους λένε όχι ε, και όταν θέλουν να θέσουν ένα ερώτημα δεν δέχεται ο άλλος το ερώτημα. Η Ευρώπη μας παρακολουθεί. Η κρίση την οποία ζούμε υπάρχει σε όλες τις χώρες. Υπάρχει και στη Γερμανία. Η στήριξη των δύο μεγάλων κομμάτων έχει μειωθεί και παρά έναν πρόεδρο ο οποίος στη Γαλλία τον θαυμάζει όλη η Ευρώπη δεν τον θαυμάζουν οι πολίτες του. Αν πράγματι θέλουμε να υπερασπιστούμε την ευρωπαϊκή συνεργασία, αν πράγματι θέλουμε η Ευρώπη να συνεχίσει να υπάρχει, θα πρέπει να αλλάξουμε τις πολιτικές μας, γιατί η πολιτική μας απειλεί και απειλήσε τους Βρετανούς. Μετανάστευση, ευρωπαϊκό στρατός, κοινό νόμισμα, αν τα αλλάξουμε όλα αυτά τότε θα αλλάξουμε σωστά την Ευρώπη. Ο κύριος Χατζηγεωργίου για ένα λεπτό. Έχει δώσει κατεύθυνση προς το Βουλή των Κοινοτήτων για επαναπροβληματισμό και νομίζω ότι και εγώ γενικά πράγματα μπορεί να πω. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα ψες δεν ήταν ήττα της Βρετανικής κυβέρνησης μόνον, ήταν ήττα κατά την άποψή μου της μεγαλαυχίας των πολιτικών εξουσιών διαχρονικά και βεβαίως της βρετανικής μεγαλαυχίας διαχρονικά. Δεύτερο, πρέπει να κάνουμε αναφορά σήμερα σε ένα όνομα ένα και του οποίου βρισκόμαστε σήμερα εδώ και ένα και του οποίου βρίσκεται ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία σε αυτήν την κατάσταση. Και είναι το όνομα του κυρίου David Cameron. Γιατί το λέω, όχι για να χλεβάσω, αλλά για να πω ότι οι μεγάλοι ηγέτες στις κρίσιμες ώρες δεν κάνουν παιχνίδια δεν παίζουμε χαρτοπέγνιο δεν είμαστε γκάμπλερς. το τρίτο δημοψηφίσματα πρέπει να γίνονται με φιδό ιδιαίτερα όταν οι σημερινοί αποφασίζουν για το πώς θα ζουν εδώ οι άνθρωποι έναν αιώνα μετά. Με φιδό τα δημοψηφίσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολλά αρνητικά πράγματα συμβαίνουν. Αυτό είναι άσχημο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον Ομένο Βασίλειο. Συμφωνώ. Οι, οι Βρετανοί εκλογείς ε, παρεπλανήθησαν μέσω ψεμάτων. Τώρα πληρώνουμε το τίμημα στον λαϊκισμό. Τώρα ε, γνωρίζουμε τι σημαίνει μια συμφωνία. Τι έχουμε ενώπιον μας, ε, ή να αποχωρήσουν χωρίς συμφωνία ή παραμονή. Να αποφασίσει ο λαός. Πολλές επιχειρήσεις εγκαταλείπουν το Ηνωμένο Βασίλειο και πολλοί Βρετανοί πολίτες ζητούν ε, υπηκότητα άλλης χώρας της Ένωσης. Εγώ είμαι υπέρ περισσότερης Ευρώπης. Ήθελα να απαντήσω στον κύριο Καμάλ, επικεφαλής των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών και στον κύριο Φάρατζαλ. αλλά έφυγαν, έφυγαν και οι δύο. Βεβαίω. Δεν του ενδιαφέρει η συζήτηση, μόνο να μιλήσουν. Ο Ντέιβιτ Κάμερον έχει την ευθύνη του Brexit, διότι ζήτησε ε, από το λαό να ψηφίσει. Ήθελε να επεκληγεί βεβαίω. Θα ήθελα να χαιρετήσω, να συγχαρώ τον Μισελ Μπαρνιέ και την ομάδα του, διότι δικαίω λέει ότι αυτή η συμφωνία των 600 σελίδων είναι ο καλύτερος δυνατός συμβιβασμός. Και βεβαίω το πρόβλημα θα παραφράσω την Μάργαρετ Θράτσετ νομίζω ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Η μόνη εναλλακτική είναι η χαοτική ε, κατάσταση σήμερα. Θα μπορούσε να δώσει χρόνο στο χρόνο και στο επίπεδο του Ηνωμένου Βασιλείου. Νομίζω ότι πέραν από τους λαϊκιστές ε, είναι η λογική ε, που θα υπερισχύσουν διότι έχουμε όλοι συμφέρον να παραμείνει. Δεν θα υπάρξει Brexit. Το κύριος Στάμπατ. κυρία Πρόεδρε. Ξέρουμε ότι απέτυχε η συμφωνία που ήταν επιτάπητος. Οπότε ή θα υπάρξει ένα καταστροφικό Brexit που θα δημιουργήσει προβλήματα και στη Βόρεια Ιρλανδία. Οπότε το μόνο που μένει είναι να ρωτήσουμε το λαό. Αλλά βεβαίως ορισμένοι λένε μα τους ρωτήσαμε ήδη. Δεν είναι δημοκρατικό να τους ξαναρωτήσουμε. Αλλά η δημοκρατία είναι η κυριαρχία του λαού και δεν χρειάζεται να επιμείνουμε σε ένα λάθο. Το καλύτερο θα ήταν να ξαναρωτηθεί ο λαός με το ερώτημα. Θέλετε σε διαπραγματεύσει με τα θεσμικά όργανα να βρείτε μια άλλη λύση. Και θέλω να κάνω πραγματικά παράκληση προς το σώμα αυτό. Δεν πρέπει να διαπραγματευόμεθα υπεροπτικά. Όλα όσα άκουσα εδώ ε, είναι να τιμωρηθεί η Βρετανία. Αυτή είναι η λάθος προσέγγιση. Πρέπει να καταλάβουμε ότι χρειαζόμαστε το Ηνωμένο Βασίλειο για την Ευρώπη. Εάν γίνει έτσι συζήτηση θα καταλήξουμε θετικά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φλάναγκαν επόμενο. Το πρώτο που πρέπει να υποθεί και δεν, συμφωνεί, δεν συμφωνώ συχνά με τον Κέλλη είναι να επανέλθουμε σε αυτό που είπε η Αλίν Φώστα ότι δεν πρέπει να υπάρξουν ποτέ σκληρά σύνορα στη Βόρεια Ιρλανδία. Δεν υπήρξαν ποτέ σκληρά σύνορα. Μα πού ήταν όταν υπήρξαν ε, σκληρά σύνορα. Ίσως για εκείνη δεν, ε, δεν ε, υπήρχαν για εκείνη, αλλά είχαμε σκληρά σύνορα. Είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε παράταση του άρθρου 50. Αυτό το σκάκι που παίζεται δεν θα καταλήξει καλά. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μας εξηγήσει πώς θα βοηθήσει την Ιρλανδική οικονομία και ιδιαίτερα τους γεωργούς μας. Άκουσα ε, ένα σχόλιο από τον Κονθάλεθ Πόνς ότι δεν είναι πρόβλημα της Ευρώπης. Αλλά βεβαίως ναι, θα το δημιούργησε η Ευρώπη και αυτό το κατανοώ. Βεβαίως, αλλά όσο και να το πούμε, είναι τώρα, έχει καταστεί και δικό μας πρόβλημα. Εμείς στην Δημοκρατία της Ιρλανδίας είμαστε μέλος της Ένωσης. Μας δημιουργεί τρομερά προβλήματα η κατάσταση. Το να λέτε ότι δεν είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα λοιπόν είναι λάθος. Πρέπει να αλλάξετε στάση. Και κύριε Μπαρνιέ, Πρέπει να πω ότι ανησυχούσα στην αρχή για σας, αλλά έκανε καταπληκτική δουλειά. Συγχαρητήρια, κρατήσατε την πυκρεμία σας όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φράγκαλη, πρόεδρος. Ε, τώρα δίνω τον λόγο στον κύριο Χόκμαρκ. Κυρία Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα σχετικά με τους συναδέλφους του UKIP από ό,τι καταλαβαίνω δεν έχουν ούτε μία έδρα στο Westminster. Καμία έδρα εκλεγμένη από τον λαό της Μεγάλης Βρετανίας για να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν το μέλλον του Ηνωμένου Βασιλείου. Και νομίζω ότι έχει σημασία αυτό. Αλλά επίσης ο κύριος ε, Φαράτζ, θα ήσασταν ευγνώμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είχατε καμία αντιπροσώπευση κοινοβουλευτική, πουθενά. Δεύτερο, σχετικά με τους Βρετανούς φίλους μας ε, και με αυτούς που ασχολούνται με το θέμα στο Westminster. Αν θέλουν παράταση, χρόνο για προβληματισμό, αν θέλουν να επανέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήθελαμε να τους πούμε ότι είναι πρόσδεκτοι. Και η κυρία Γραπίνη τώρα. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Πάρα πολλά πράγματα λέχθηκαν εδώ. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ ε, σημαντικό. Βλέπουμε ότι υπάρχει πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θέλει το Ηνωμένο Βασίλειο να παραμείνει μεταξύ μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον διαπραγματευτή. Το πρόβλημα δεν δικό μας, αλλά είναι πρόβλημα της Μεγάλης Βρετανίας ε, και θέλω ε, το, να δούμε τι θα γίνει με το μέλλον ε, των πολιτών μας που ζουν εκεί και αυτών της Μεγάλης Βρετανίας που ζουν εδώ. Το μέλλον το εμπορικό. Όχι μόνο πρέπει να συνεχίσουμε τη διαπραγμάτευση, αλλά θα πρέπει και ο πληθυσμός, ο οποίος στην πλειοψηφία του θέλει να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πήγα στο Λονδίνο, στο Μπέρμιγκα, μίλησα με τους πολίτες, με τους επιχειρηματίες. Θέλουν ε, να παραμείνουν. Είναι οι πολιτικοί άνδρες που δίνουν την κατεύθυνση αυτή της δεξιάς που ε, ρίχνουν μηνύματα που λένε ότι αν βγει το Ηνωμένο Βασίλειο ε, θα πληρώνουμε εμείς τις συντάξεις στους Μεγάλους Βρετανούς. Ωραία, τώρα ολοκληρώνω τη διαδικασία στη του και δίνω το λόγο στον Αντιπρόεδρο κύριο Τίμερμαντ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε χωρίς ε, την συμπαράσταση των Βρετανών στην ε, πιο δυσχερή και πιο ζωφερή στιγμή της ιστορίας μας δεν θα ήμασταν εδώ μέσα αυτή τη στιγμή. Και η δική μου χώρα ε, είναι ευγνώμων για την ελευθερία που μας έδωσαν οι Βρετανοί στρατιώτες. Είναι άρρηκτη η δεσμή μεταξύ της Βρετανίας και της Ευρώπης. Είτε είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε όχι. Πάντα θα είναι τμήμα της Ευρώπης η Βρετανία. Με έναν τρόπο που θα καθορίζει το κοινό μας πεπρωμένο και λυπάμαι που βλέπω να είναι τόσο διηρημένο όσο σήμερα το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι διαιρέσεις που έχουν, που προκληθεί από τον Brexit έχουν παραλύσει την Βρετανική κοινωνία. Εγώ θα παραμείνω αιώνια ευγνώμων. Όχι μόνο για την ελευθερία μας, αλλά και για τους Βρετανούς ε, δασκάλους που είχα όταν ήμουν νέος, που μου έμαθαν να αγαπώ τη Βρετανική λογοτεχνία, την τέχνη, μου έμαθαν τη γλώσσα, αυτό δεν θα αλλάξει ό,τι και να συμβεί. Αλλά θέλω να καταστήσω κάτι απόλυτα σαφέ, αντιδρώντα ορισμένα που ελέγχθησαν από τον κύριο Καμάλ και τον κύριο Φαράτζ. Εγώ στην Επιτροπή με τον Μισελ, ούτε σε καμία από τις 27 πρωτεύουσε δεν διαπίστωσα καμία τιμωρητική διάθεση σε αυτή τη διαδικασία. Κανεί δεν θέλει να τιμωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο που αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. στις διαπραγματεύσεις σε όλες τις πρωτεύουσες και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η στάση μας ήταν να γίνει η μικρότερη δυνατή βλάβη σε αυτή τη διαδικασία αλλά να μην αυταπατώμεθα ζημιά θα γίνει το Brexit θα κάνει ζημιά στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η κοινή μας ευθύνη να περιορίσουμε αυτή τη βλάβη όσο γίνεται Τι θα γίνει τώρα στις επόμενες εβδομάδες, μήνες, ίσω και χρόνια. αυτό θα το αποφασίσει ο Βρετανικός λαός. Και πρώτα απ' όλα η Βουλή των Κοινοτήτων, όπου θα γίνουν οι συζητήσεις. Εμείς ε, θα παίξουμε το παιχνίδι όπως θα καθορίσει ε, το Ηνωμένο Βασίλειο πώς θα παιχθεί περαιτέρω. Ε, ποτέ δεν έκρυψα. Θα προτιμούσα να παραμείνει η ε, Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό εξαρτάται από του Βρετανού πολιτικού, όχι από εμά. Και κάτι που θέλω επίση να καταστήσω σαφέ, ε, επειδή άκουσα τον κύριο Καμάλ που είπε ότι υπάρχει ενή αγορά και άλλα στοιχεία. Αλλά δεν μπορεί κανεί να πει θα φύγω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα κρατήσω όλα τα στοιχεία που μου αρέσουν χωρί να καταλαβαίνει πώ θίγει αυτό την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί ω Ευρωπαίοι πολιτικοί, ω κράτη-μέλη, ω θεσμοί, έχουμε υποχρέωση να διασφαλίσουμε το ουσιώδη στοιχεία του τι σημαίνει να είναι κανείς μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το αδιέρετο των τεσσάρων ελευθεριών. Είναι η ακαιρεότητα τη ενιάία αγοράς. Αυτά είναι αδιαπραγμάτευτα. Κάτι που με καταπλήσει επίσης. Είναι ότι ο κύριος Φάρατζ έχει αυτό το όνειρο, το ψευδές όνειρο περί ανεξαρτησίας που τον οδηγεί στο να αγνοεί εντελώ τη θεμελιώδη σημασία τη Συμφωνία τη Μεγάλη Παρασκευή για την ειρήνη στην Ευρώπη. Είναι απόλυτα σαφέ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχουμε συλλογική ευθύνη ως Ευρωπαίοι να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνει η ειρήνη στο νησί της Ιρλανδίας. Και με βάση την ανάλυση μας. Για να υπάρξει αυτή η ειρήνη δεν πρέπει να υπάρχουν σκληρά σύνορα στο νησί της Ιρλανδίας. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε τον backstop. Και αυτό είναι διαπραγματευτό. Και πραγματικά τρελαίνεται ο άνθρωπος όταν ε, από τη μία βλέπει να υπάρχει τέτοια ευρωπαϊκή αλληλεγγύη που κανείς στις 27 ε, ε, πρωτεύουσες λέει ε, δεν θεωρεί ότι μπορούμε να καταλήψουμε την Ιρλανδία. Και πολλοί στο Westminster δεν βλέπουν την ουσιώδη αξία της Συμφωνίας Μεγάλης Παρασκευής. Και γι' αυτό το όνειρο της υποτιθέμενης ανεξαρτησίας είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν την ειρήνη στην Ιρλανδία. Και δεν μιλάω για τις δουλειές, τις επενδύσεις και όλα αυτά. Θα ήταν ειλικρινές σε αυτή την εκστρατεία που οδήγησε στην ε, απόφαση για τον Brexit, την οποία απόφαση σεβόμεθα. Θα ήταν καλό να πούνε ότι θέλουμε τόσο πολύ την ε, ελευθερία μας που δεν, θέλουμε, που δεν μας ενδιαφέρει αν θα χάσετε δουλειά για τις επενδύσεις, για το σύστημα υγείας. Δεν μας ενδιαφέρει ότι θα υπάρχουν ποτηγιαρίσματα στους δρόμους. Θέλουμε την ανεξαρτησία μας ανεξαρτήτως συνεπειών. Αυτό θα ήταν μια ειλικρινής προεκλογική εκστρατεία υπέρ του Brexit. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις στο Westminster, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα συνεχίσουμε ειλικρινά να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γίνει όσο λιγότερο μικρότερη ζημιά όπως και αν διαμορφωθεί η κατάσταση. Κύριε Καμάλ, αναφερθήκατε στους You can't always get Eagles. Εγώ θα αναφερθώ στους Rolling Stones. Δεν μπορείς πάντα να ε, αποκτήσει αυτό που θέλεις αλλά αν προσπαθήσεις αρκετά σκληρά μπορεί να αποκτήσει αυτό που χρειάζεσαι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Βεβαίω ε, ε, θα θέλαμε όλοι εδώ να έχουν την ίδια απόψη και τώρα δίνω τον λόγο στην κυρία Τσιότ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι θα πρέπει να ελπίζουμε ότι οι βουλευτές στο Ηνωμένο Βασίλειο θα οδηγήσουν σε ένα αποτέλεσμα που θα οδηγήσει ε, σε συντεταγμένη έξοδο και θα πρέπει να υποστηρίξουμε μια τέτοια διαδικασία. Εάν αυτό το θετικό σενάριο υλοποιηθεί, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι η συμφωνία της 25ης Νοεμβρίου ήταν το πρώτο βήμα σε μια μακρά διαδικασία θα πρέπει η εφαρμογή ε, του Συμφωνίας Αποχώρησης να παρακολουθείται στενά, ούτω